Dear colleagues, welcome to the Budgets Committee meeting. Κυρίες και κύριοι, καλώ ήρθατε στη συνεδρία τη Επιτροπή Προπολογισμών. Πρώτο σημείο είναι η έγκριση της ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται. Δεύτερο σημείο, ανακοινώσει του Προέδρου. Μετά από τη γραπτή διαδικασία, τις γραπτές διαδικασίες μάλλον, που ακολουθήθηκαν οι συντονιστέ αποφάσισαν να συντάξουν έκθεση θέματα έκτακτα μέτρα ε, όσον αφορά το Brexit. Και υπάρχει κανονισμός του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή, ε, την υλοποίηση του προπολογισμού του 2019 και να λάβουμε υπόψη και την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η για το θέμα αυτό θα είναι ο πρόεδρος μας, ο κ. Αχτουή. Δεύτερο, οι συντονιστές αποφάσισαν να συντάξουν γνωμοδότηση υπό τη μορφή επιστολής προς την Επιτροπή Ρέτζη έκθεση για τους πόρους, για τη συγκεκριμένη ε, πρικοδότηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των ε, νέων. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις ανακοινώσεις, έγκριση των πρακτικών της συνεδριάσεως της 23ης Ιανουαρίου δεν υπήρχαν ενστάσεις και αντιρρήσεις. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Και πάμε στις ψηφοφορίες. Καταρχήν, κεφάλαιο 3 προπολογισμού του 2019, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπάρχουν αιτήσει για μεταφορές κονδυλίων. Θεωρούμε ότι έχει λήξει αυτό το θέμα. Σημείο 5. το άλλη τομή του προβλησμού 2019. Τον κύριο Ρούμπικ έχουμε τον εισηγητή και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά. Σαν αφορά τα άλλα τμήματα, υπάρχουν δύο αιτήσει για μεταφορές. Η μία προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το ευρώ στο σημερινό προϋπολογισμό πρέπει να μεταφερθούν και πρόκειται για την γραμμή 227 δαπάνες ε, για έντυπο υλικό, έγγραφα κτλ. Πιστεύω ότι δικαιολογούνται αυτές οι μεταφορές, αυτό το ποσό. Και η δεύτερη αίτηση είναι από την Επιτροπή των Περιφερειών, 200.000 ευρώ για τον προϋπολογισμό που ουσιαστικά καλύπτει τα έξοδα επικοινωνίας ε, για τις πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι και αυτό είναι λογικό και δικαιολογείται. Η Επιτροπή των Περιφερειών επίσης ε, συμμετέχει στις ευρωπαϊκές εκλογές, ε, στηρίζει την δημοκρατία και νομίζω ότι πρέπει να εγκρίνουμε τα ποσά αυτά που μας ζητάνε. Σας ευχαριστώ κύριε Ρούμπικ. Οι σκιώδεις επιθυμούν να ομιλήσουν. Η κυρία Καρουαζαμπάλ από τους σοσιαλιστές. Άλλος δεν υπάρχει. Αφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, οι μεταφορές θεωρούν ως, θεωρούνται εγκεκριμένε. Εγκρίνονται λοιπόν. Σημείο 6. Ε, η πολιτική για τα κτίρια. Δεν λάβαμε κάποιο αίτημα. Σημείο 7. Η πολιτική λοιπόν για τα κτίρια. Δεν έχουμε νέες ε, πληροφορίες. Η κυρία Χολμάιρα απουσιάζει σήμερα. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Σημείο 8. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προπολογισμό του 2020 κεφάλαιο 3 τμήμα 3. Έχουμε 114 τροπολογίες προς εξέταση. 114 υπερλήφθανε για το σχέδιο προσανατολισμών για τον προπολογισμό του 2020. Η κυρία Χολμάιερ λοιπόν είναι υπεύθυνη, δεν είναι παρούσα και ο κύριος Ρούμπικ θα την αντικαταστήσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά. Δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα η κυρία Χολμάιερ αλλά έχει καταθέσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα. Και εστιάζει τη δουλειά της στην επεξεργασία των ε, συμβιβαστικών. Έχουμε περίπου 140 τροπολογίες, κυρίως για την έρευνα και την ε, ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος, καταπολέμηση της ενεργείας ιδίως των νέων, ψηφιοποίηση, ασφάλεια ε, και στελέχωση των εκτελεστικών οργανισμών. Ο στόχος είναι να είναι ο προεπλησμός του 2020 γέφυρα για το επόμενο μισονομικό πλαίσιο και ξέρουμε ότι υπάρχουν οι διαβουλεύσεις που γίνονται και θα πρέπει και εμείς να παράσχουμε την άποψή μας για ένα μακροπρόθεσμο όραμα που θα επιτρέψει την εκπλήρωση των στόχων της Ένωσης. Το 2020 είναι βάση για την επόμενη επταετία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Η στρατηγική που θέλει να προτείνει η κυρία Χολμάιερ είναι να αξιοποιήσουμε όλη την ευελιξία του δημοσιονομικού πλαισίου, πάντοτε το τόνιζε αυτό, και να ληφθούν όλα τα ε, σχετικά μέτρα, να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες προσφέρει ο προπολογισμό, έρευνα καινοτομία, θέλουμε τον ορίζοντα 2020 να τον ενισχύσουμε. Τα τελευταία πέντε χρόνια ε, πάντα αυτή ήταν η θέση μας και ήταν και η δύναμη, αν θέλετε, της Ένωσης, για βασικές τεχνολογίες ε, και η κυρία ε, Χολμάιερ θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε κάθετοι. Επίσης ε, πλήρω ε, μεταφορές, γεωργία, μεταξύ άλλων θα παίξουν σημαντικό ρόλο και στο μέλλον και ψηφιοποίηση επίσης, ε, ο σημαντικός ρόλος της ψηφιοποίησης, ο μετασχηματισμός, ε, πρέπει να στηρίξουμε το μετασχηματισμό της οικονομίας και βέβαια προσέγγιση ε, στους πολίτες, κατάρτιση και ψηφιακές δεξιότητες και κυβερνοασφάλεια και άμυνα στον κυβερνοχώρο, το ψηφιακή Ευρώπη, το Connecting Europe, θα παίξουν αυτά τα μέσα σημαντικό ρόλο αν θέλουμε η Ένωση να είναι ανεξάρτητη και να μπορέσει να στηρίξει και την ε, στρατηγική της εκεί. Επίσης, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, προστασία εξωτερικών συνόρων, αλλά και εσωτερική ασφάλεια, εντός ενώσης ε, θέλουμε κατάργηση των ε, ελέγχων, στα εσωτερικά δηλαδή σύνορα, αλλά θέλουμε τη βέλτιστη δυνατή προστασία στα σύνορα. Άρα ασφάλεια, δικαιοσύνη, μετανάστευση, άσυλο και φορεί σχετική, εκεί θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση και το απαραίτητο προσωπικό. Ε, δεν είμαστε πολύ ευέλικτοι, δεν μπορούμε να διαθέσουμε υπερβολικούς πόρους και μέσα. Ξέρουμε ότι τα τελευταία 15 χρόνια από το 1,2 του ΑΕΠ έπεσε στο 0,9% ε, του ΑΕΠ ε, ο προπολογισμό και άρα μειώνονται τα περιθώρια για τη χρηματοδότηση και στην επόμενη επταετία. Εξού και πόσο σημαντικό είναι να συντονίσουμε σωστά τις ε, διάφορες δραστηριότητες ώστε το θέμα κυβερνοσφάλεια, ασφάλεια από απειλέ στον κυβερνοχώρο, ψευδή ειδήσει, παραπληροφόρηση, πρέπει σε αυτού του τομεί να έχουμε παρκή χρηματοδότηση. Ιδίω όταν μιλάμε για επιθέσει εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα σημαντικό μέλημα. Η Ευρώπη από κοινού θα πρέπει να καταπολεμήσει το πρόβλημα της παραπληροφόρησης. Και αυτό ε, και εν ώψη των ευρωεκλογών, για να περάσουμε αυτό το μήνυμα στους πολίτες. Υπάρχει συνένεση ε, σαφής νομίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας ε, στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ε, γιατί αυτό μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Μπορεί να αποτελέσει προστέμενη αξία και για τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Και νομίζω το κόστος της μη Ευρώπης ιδίως για τα ασθενή κοινωνικά στρώματα ε, είναι σαφές και γι' αυτό νομίζω ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα. Επίσης, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αλληλεγγύη στην Ευρώπη, στις τελευταίες διαβουλεύσεις, πραγματεύσει ε, καταδείξαμε πόσο σημαντικό είναι το Erasmus Plus ε, ως πρόγραμμα ιδίως για τους νέους και για τους σπουδαστέ και από τα διάφορα κοινωνικά στρώματα και υπόβαθρα. Είναι σημαντικό και τη Youth Employment Initiative, αυτή την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, ε, να κάνουμε και το 19 και το 20 αυτή την πρωτοβουλία επιτυχία για εμείς θέλαμε πιο πολλά χρήματα, 370 εκατομμύρια και 205 εκατομμύρια για την έρευνα, τα πρώτα για το Εράσμο. Ένα δις ε, θέλουμε να διατεθεί συνολικά για όλα αυτά τα προγράμματα. για να έχουν μια ομαλή μετάβαση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Σε ό,τι αφορά τώρα την μακροπρόθεσμη λύση που πρέπει να βρεθεί στο μεταναστευτικό φαινόμενο και εκεί συμφωνούμε γιατί έχει οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές επιπτώσεις επέπφυσκα να στηρίξουμε τα κράτη, με μετερικές σχέσεις, ιδίως με τις χώρες Αφρικανικής Υπήρου. Η στόχη βιώσιμη ανάπτυξη επίση είναι κάτι σημαντικό, ιδίω ο δεύτερο στόχος που είναι ασφαλή τρόφιμα, βιώσιμα τρόφιμα. Το 6 για, για υδροδότηση αποχέτευση και το 7 ανανεώσιμες πηγές. Ιδίω στην Ήπεθρο, στις λιγότερες, ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, η ανεξάρτητη ε, μάλλον η αυτονομία στην παραγωγή ενέργειας, στον εφοδιασμό σε ενέργεια είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μπορούμε να επενδύσουμε, παραδείγματος στην ολική ενέργεια και στην ηλιακή ενέργεια που υπάρχει πολύ ηλιοφάνεια. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κλιματικά ζητήματα, φυσικά και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε πιο αποφασιστικά αυτά τα ζητήματα. Θέλουμε να είμαστε πρωτοποριακοί και στην κυκλική οικονομία και επίσης ε, θέλουμε μια πλευρά πλευράς κλίματος ουδέτερη ε, βιομηχανία και κοινωνία. Θέλουμε περισσότερη παραγωγή πίσω στην Ευρώπη από εταιρείε που έχουμε εγκατασταθεί εκτό. Θέλουμε λοιπόν μια πιο ελκυστική Ευρώπη και θέλουμε να προσελκύσουμε επενδύσει για να έχουμε και νέε θέσει εργασία με καλέ αποδοχέ. Αυτό είναι επίση κάτι πολύ σημαντικό. Και από τη ρομποτική, το τεχνητή νοημοσύνη, τη βιομηχανία 4.0 μπορούμε με όλα αυτά να μιλήσουμε νέε θέσει εργασία. Ε, ε, όλο αυτό για μένα είναι ένα σχέδιο προς απασχόλησης και μπορούμε να συνεισφέρουμε. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατάρτιση του προπολογισμού το 2020, θα ακολουθήσουμε την ίδια γραμμή με το 19, δηλαδή θέλουμε το 15.3 άρθρο να εφαρμοστεί. Πρέπει να υπάρξει μεταφορά αυτών των πιστώσεων από το Συμβούλιο, είτε είναι περισσότερο είτε είναι λιγότερα. Πρέπει επίση η Κομισιόν να μα ενημερώσει για το ποσοστό των ε, μεταφορών αυτών και της αποδέσμευσης των κονδυλίων, τα λεγόμενα decommitments. Έτσι θα έχουμε, πιστεύω, και τη δυνατότητα να δημορφώσουμε ένα συνεκτικό επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Η βάση για αυτό, παραλαμβάνω, είναι το προπολογισμό του 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Ρούμπικ. Οι σκιώδεις η κυρία Μωράν για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, όπως μας υπενθύμησε ο κύριος Ρουμπίχ και ακριβώς επειδή υπήρχαν συνομιλίες με την κυρία Χολμάιερ, σας επιβεβαιώνω και αποσαφηνίζω ότι υπάρχει μεγάλη σύγκληση μεταξύ των ε, θέσεων που εκφράζουν οι τροπολογίες. Βεβαίως ο προϋπολογισμός του 2020 θα πρέπει να αποτελέσει γέφυρα προς το επόμενο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει ο προϋπολογισμός του 2020 να έχει δυνατότητες γιατί είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός του πολιετούς δημοσιονομικού προγράμματος να μπορεί λοιπόν να έχει τη δυνατότητα να αποφύγει και να εξουδετερώσει κρίσεις. Όπως υπενθύμησε ο κύριος Ρουιμπίκ, το Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να επιβεβαιώσει ένα φιλόδοξο προϋπολογισμό που ουσιαστικά στηρίζει την έρευνα, την καινοτομία, την ε, ενεργειακή μετάβαση, την ενσωμάτιση των ε, προσφύγων, το θέμα της ψηφιακής ε, σύνδεσης και βεβαίως μια σημαντική στήριξη προς τους νέους. Μέσω προγραμμάτων όπως το Εράσμους που το 2019 αποτέλεσε μια σημαντική συνιστόσα του προϋπολογισμού μας. Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις, κοινωνικές, οικονομικές, που αντιμετωπίζουμε σήμερα για μια κοινωνία η οποία δεν θα οδηγήσει αποκλεισμούς. Θέλω να σας υπενθυμίσω και τέσσερα σημεία, τα οποία βεβαίως ε, αποτελούν αντικείμενα συζήτησης, αλλά επικοδομητική συζήτησης, τη χρήση όλων των δυνατοτήτων ευελιξίας για να υπάρξει μια σταθερή χρηματοδότηση αυτού του προϋπολογισμού, άρθρο 15.3 του Μοζονικού Κανονισμού που υπενθυμίσατε. Δεύτερον, η χρήση όλων των εργαλείων που επιτρέπει ο παρόν προϋπολογισμός για την υλοποίηση όλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως τους ε, διατυπώνει ο Χάρης Εθνών για την καταπολέμηση των κλιματικών προκλήσεων εν ώψη των ε, στόχων του Παρισιού. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι η ασφάλεια και η μετανάστευση, χωρίς να υπάρχει σύγχυση μεταξύ αυτών των δύο θεμάτων και βεβαίως ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. Ενίσχυση των προϋπολογισμών της Frontex, της Europol, κάτι το απαραίτητο, και την ίδια ώρα η ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μία από τις βάσεις της ενσωμάτωσης και της ολοκλήρωσης. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση λοιπόν να υπάρχει σύγχυση μεταξύ αυτών των δύο στόχων. Κύριε Ρούμπικ, υπενθυμίσατε την ενίσχυση ή τουλάχιστον την διατήρηση των ποσών που αφορούν τις πρωτοβουλίες για την απασχόληση των νέων. Αυτό είναι καθοριστικό για το 2020 και είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Επιτροπής μας, αλλά και εμάς. Ήταν στην καρδιά των διαπραγματεύσεων το θέμα αυτό. Υπήρχαν κάποιες ε, κριτικές για το θέμα αυτό, αλλά σήμερα βλέπουμε ότι η κατανάλωση αυτών των κονδυλίων είναι σωστή, πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις δυνατότητες που προσφέρουμε στους νέους για κατάρτιση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να συνεχίσουν να στηρίζουν και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει τα ευρωπαϊκά κονδύλια να αντικαταστήσουν τα εθνικά για αυτό το σκοπό. Αυτά είναι τα τέσσερα για μένα σημαντικά σημεία. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι πριν υποβληθούν οι τροπολογίες είχαμε πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση και ελπίζω η έκθεση αυτή για τον προϋπολογισμό του 2020 θα συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας με τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Δεν βλέπω εκπρόσωπο του ECR παρόντα. Ο κ. Ντεπρέ από την Άλντε θέλει να μιλήσει εκ μέρους του κ. Τόλβαλτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν ήθελα να μιλήσω, δεν προβλεπόταν. Αλλά ο σκιώδης ηγητής του Άλντε, ο Νίλς Τόρβαλτ, δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραστεί και μου ζήτησε να παρουσιάσει τα σχόλιά του. Εν πρώτης, επιθυμεί και ευχαριστώ την κυρία Αλμάιρ για τη δουλειά που έκανε και για την έξοχη συνεργασία που ξεκίνησε με τον σκιώδη συγητή στην προετοιμασία των προσανατολισμών αυτών για τον προϋπολογισμό του 2020. Ο φίλος μας ο Τόρβαλτς θεωρεί ότι οι συμβαστικές λύσεις που δέχτηκε η κυρία Ολμάιρ είναι έξοχη αφετηρία αφετηρίες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με το Συμβούλιο. Επιμένει και επιμένω κι εγώ επί αναγκαιότητα ενίσχυση ενίσχυσης της δράσης κατά της αλλαγής του κλίματος, της θέρμανσης του πλανήτη. Ήδη τοποθετηθήκαμε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων του προπολογισμού του 2019. Είπαμε ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν σέβεται τι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει όσον αφορά ε, τη διάρκεια της περίοδου των μέτρων 2014-2020, 20% των πιστώσεων θα διατίθενται για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και για την προστασία ε, του ε, του περιβάλλοντος. Για το 2020 η πρώτη της Ευρωπαϊκής σέβεται το 20%. Αλλά αν δούμε το άθροισμα του ποσού για όλη την περίοδο δεν φτάνουμε στο 20% κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε σοβαρή προσπάθεια στα πλαίσια του προπολογισμού του 2020, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους. Εκτιμούμε το ότι τονίζει η κυρία Ολμάιρ την έρευνα, την καινοτομία, καθώς και την ανάπτυξη των ΜΜΕ, των μικρομεσών επιχειρήσεων. Έχουμε, δεχτεί, έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά το άσυλο. Αυτό θέλουμε να τονίσουμε. Είναι σημαντικό να διατίθενται περισσότεροι πόροι για την καταπολέμηση των αιτίων τη μετανάστευση. Μετανάστευση που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Πρέπει να ενισχύσουμε τα μέσα που επιτρέπουν αποτελεσματικότερα τον έλεγχο των συνόρων, να βελτιωθεί η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και πρέπει να καταπολεμηθεί η κυβερνοεγκληματικότητα. Ο κ. Τόρβαλς πιστεύει επίσης ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία από ό,τι τώρα στην καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων τις απόπειρες παραπληροφόρηση που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια και τώρα γίνονται και θα ενισχυθούν στο μέλλον ενώπιον των ευρωεκλογών. Ο κ. Πούτιν, σύμφωνα με τι συμφωνίε που κυκλοφορούν από ό,τι λένε, ενδιαφέρονται πολύ τι εργασίε μα. Το λέω εν είδη ανεκδότο διότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα μας δείχνουν ότι ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν, η κυρία Ελίζα Βέτα Πέσκοβα, η εκπρόσωπος του, είναι σταζιέρ ενός ευρωβουλευτού. Δεν ξέρω αν αυτό να μας κάνει να γελάσουμε, να ενδιαφερθούμε, αλλά ήθελα εδώ κλείνοντας την παρέμβασή μου αυτό να το αναφέρω. want to um, maybe make a note to all of you that she doesn't seem to be present in this meeting anyway. Κοιτάξτε, δεν είναι παρόν, παρούσα σε αυτή τη συνεδρία τουλάχιστον. Ο κ. Σολέ για τους πρασίνους έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Τα συζητήσαμε αυτά στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τους προσανατολισμούς η ομάδα μου υπέβαλε έξι τροπολογίες. Εστιαζόταν κυρίως στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, βιώσιμης προστασίας του περιβάλλοντος, να μην βασίζεται η οικονομία μας στον άνθρακα, δυνάμει, συμφωνιών που έχουμε συνάψει, όπως είπε και ο κ. Ντεπρέ, Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολείπεται των στόχων για το κλίμα, στόχων που είχαν τεθεί για το τέλος του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου, θα έχουμε αποτύχει έτσι που πάμε. Άρα πρέπει να αυξήσουμε τις δαπάνες για το κλίμα. Πρέπει επίσης η διάσταση του κλίματος να λαμβάνει υπόψη σε όλες τις πολιτικές. Στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών, της γεωργίας, Αυτό είναι ο βασικό στόχο των τροπολογιών που αποβάλαμε. Έχουμε και άλλε ανησυχίε. Οι περισσότερε αναφέρθηκαν από του συναδέλφου. Εν πάση περιπτώσει, προσβλέπω στι συνομιλίε που θα λάβουν χώρα βάσει των συμβαστικών που θα ετοιμάσει η συγκήτρια. Ευχαριστώ. Γκουε, δεν υπάρχει κάποιο. Άλλο που ενδιαφέρεται να μιλήσει για το θέμα αυτό, όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως έχει κάτι να πει. Ορίστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την πλευρά μας ευπρόσδεκτη ανταλλαγή απόψεων. Όπως ήδη διαφάνει από την προηγούμενη συνεδρίαση και που παγιώθηκε και εδώ αυτή η άποψη υπάρχει μεγάλη σύγκληση όσον αφορά τις προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Αυτό είναι καλό. Να επενθυμίσω κάτι ότι όσον αφορά τι αναλήψει υποχρεώσεων, όπως ήδη ίσχυσε και τα προηγούμενα χρόνια, πιθανότατα και το 2020 θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολύ τα μέσα ευελιξίας για τη χρηματοδότηση ε, των υποχρεώσεων αυτών, κυρίως στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας, αλλά και για τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Σε μεγάλο βαθμό Χάρη στη συμπληρωματική ευελιξία που πέτυχε το Κοινοβούλιο σε πρώτε διαπραγματεύσει, θα έχουμε επαρκή ευελιξία για τη χρηματοδότηση των πρόσθετων αυτών αναγκών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε, όσον αφορά τι πληρωμές τη σημασία που η Επιτροπή σα στο σχέδιο προσανατολισμών θέλει να δώσει για την ενδεδειγμένη χρηματοδότηση ε, για, τις, για τους διάφορους στόχους, για τις πληρωμές. Έχουμε κοινή προσέγγιση και στο σχέδιο προπολογισμού την άνοιξη αργότερα θα δώσουμε μια σχετική πρόταση που θα είναι σωστή όσον αφορά τα ποσά. Κλείνοντας, σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπουμε σε επικοδομητικό διάλογο για τις προτεραιότητες του 2020, κυρίως κατά τον εαρινό τριμερή διάλογο του επομένου μήνα και ο Επίτροπος Έτιγκερ θα έχει περισσότερα σχόλια, με βέβαιο, όσον αφορά τι κατευθυντήριε γραμμέ και, και του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και προσβλέπουμε στη συνεργασία μα κατά τη διάρκεια όλη τη διαδικασία του προπολογισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα τελικά σα σχόλια. Ο κ. Ρούμπικ, που εκπροσωπεί την κυρία Χολμάιερ, θέλει να μιλήσει. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τις τοποθετήσεις σας. Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα σχόλιά σας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Σας παρακαλώ, θα πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, γιατί το θέμα του Brexit φυσικά θα παίξει καθοριστικό ρόλο και μέχρι την τελευταία στιγμή θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξουμε ευελιξία, γιατί όπως ξέρετε τα γεγονότα εξελίσσονται με ραγδαίο τρόπο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει για όλα αυτά τα θέματα να ψηφίσουμε όπως έχει προγραμματιστεί πριν την ολοκλήρωση της θητείας μας και πριν το νέο κοινοβούλιο συσταθεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε εμείς να επεξεργαστούμε όλες τις εναλλακτικές Ελπίζω ότι η διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και το γνωρίζω μάλλον θα είναι εξαιρετικά συναρπαστική και ενδιαφέρουσα. Thank you. Σας ευχαριστώ κύριε Ρούμπικ για το χρονοδιάγραμμα λαμβάνοντας υπόψη και το Brexit θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών 7 Μαρτίου και στην Ολομέλεια η ψηφοφορία θα γίνει στην πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου και ο παραδοσιακός το ημερής διάλογος με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει χώρα στις 20 Μαρτίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά μας. Για τον προϋπολογισμό του 2020, για τις κατευθύνσεις γραμμές του προϋπολογισμού του 2020. Στο σημείο 9 τώρα, το σημείο 9 αφορά συζήτηση με πέντε γενικές διευθύνσεις και ανταλλαγή απόψεων με αυτές, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε παρούσες γενικές διευθύνσεις. Καμία δεν είναι εδώ. Και Είχαμε πει ότι στις 3.30 θα το συζητούσαμε το θέμα ενδεικτικά. Τι να κάνουμε σας τώρα. Γιατί αν σας αφήσω να φύγετε τώρα, πού να σας μαζέψω. Θα διακόψουμε για ένα τέταρτο και θα ξαναμαζέψω το κοπάδι εδώ γύρω στις 3 και 20. Και αναμένονται γενικές διευθύνσεις ότι θα είναι εκεί, θα έχουν φτάσει τότε. Λοιπόν, ένα τέταρτο διάλειμμα.

Ευχαριστώ feel Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συνεδρία τη Επιτροπή Προπολογισμών. Είμαστε στο σημείο 9, κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020, τμήμα 1, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέρσι είχαμε μια υπέροχη εμπειρία. Είχαμε ανταλλαγή απόψεων με διάφορες γενικές διευθύνσεις για να μπορέσουμε να προβλέψουμε τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να το ξανακάνουμε, να το κάνουμε παράδοση. Αυτή τη φορά καλέψα, καλέσαμε πέντε γενικές διευθύνσεις, οι οποίες εκπροσωπούνται εδώ, έξοχη ευκαιρία για πραγματική ανταλλαγή απόψεων που θα είναι ουσιαστική με αυτές τις γενικές διευθύνσεις. Έχουμε τη Γενική διεύθυνση Inlo, Trad, Link, Fins και Inlo. Θέλουμε να δώσουμε 10 λεπτά στον καθένα, σε κάθε γενική διεύθυνση και μετά θα δώσουμε το λόγο στους κοιόδης και στα μέλη, αλλά και άλλοι μπορούν να ζητήσουν το λόγο αν επιθυμούν. Η είναι ο κύριος Μάνκα. Κύριε Μάνκα, ε, για μια σύντομη εισαγωγή σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω. Έγινε μια πρώτη συνεδρίαση των σκιωδών σήμερα. Αυτή η συνάντηση ήταν πολύ καλή κατά την άποψή μου διότι το Μάιο διεξάγονται εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε χρονική πίεση. Την Παρασκευή που δώσω την έκθεση προσχολιασμό και τη Δευτέρα όλοι θα λάβετε στα αγγλικά ένα σχέδιο εκθέσεως και έτσι μπορούμε να προετοιμάσουμε τροπολογίες για τις 7 Μαρτίου. 7 Μαρτίου θα γίνει μια παρουσίαση της έκθεσης στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών και στις 13 ε, Μαρτιού αυτή θα είναι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Θεωρητικά όλα αυτά, αλλά αυτό το πρόγραμμα θέλουμε. 25 Μαρτίου θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε τις τροπολογίες, ούτως ώστε 27 και 28 Μαρτίου στην Ολομέλεια να είμαστε θέση να εγκρίνουμε την έκθεση. Χαίρομαι που έχουμε εδώ τις γενικές διευθύνσει. Έχουμε παρόντου γενικούς διευθυντέ πέντε γενικών διευθύνσεων. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια καλή συμβολή στην συζήτησή μα. Θα σα δώσουμε το λόγο και μετά πιθανότατα θα έχω κάποιες ερωτήσεις να τους ε, απευθύνω. Ευχαριστώ κύριε Μάνκα. Πρώτη γενική διεύθυνση είναι η ΦΙΝΣ για τα οικονομικά. Ο κ. Διδιέ Κλεφή έχει το λόγο για 10 λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Μάγκια, για την πρωτοβουλία αυτή. Εκ νέου φέτος καλείται πολλές γενικές διευθύνσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε τον προϋπολογισμό μας για το 2020 με λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Όσον αφορά τη δική μας γενική διεύθυνση των οικονομικών, παρεμβαίνουμε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, είμαστε ο συντονιστής, διοικητικός συντονιστής για την προετοιμασία του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και δεύτερον, καθώς ε, είμαστε υπεύθυνοι για τις ε, δαπάνες που αφορούν τη χρηματοδότηση των πολιτικών ομάδων και χρηματοδότηση ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα καταρχήν λοιπόν να σας υπενθυμίσω ποια είναι η διαδικασία η διοικητική που φτάνουμε μέχρι το σχέδιο προϋπολογισμού της ε, Γενικές κατευθύνσεις Γραμμές. Δεύτερον, με τη δεύτερη ιδιότητά μας θα σας παρουσιάσω και τις ε, ιδιαίτερες αρμοδιότητες που έχουμε στην γενική μας διεύθυνση. Όσον αφορά την διοικητική και πολιτική διαδικασία, με έναν τρόπο που θα υπογραμμίσουμε το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε και τα αποτελέσματα των ακροάσεων Βλέπετε εδώ ότι η διαδικασία κρατάει 4 με 6 μήνες και υπάρχουν με πράσινο και με μπλε οι διάφορες διαδικασίες. Ξέρετε εξάλλου πολύ καλά ποιες είναι αυτές που ανήκουν, εμπίπτουν στη δική σας αρμοδιότητα. Το Νοέμβριο ξεκινάμε με την προετοιμασία, με συγκεκριμένες οντολές που δίνονται, ανάλυση των ε, ετοιμάτων, και κατόπιν ακρόαση για την κάθε Γενική Διεύθυνση με την Γενική Διεύθυνση των Οικονομικών. Ακολουθεί η φάση της διατησίας του Γενικού Γραμματέα δηλαδή, καθώς και η ολοκλήρωση του τελικού του εγγράφου όσον αφορά τις προβλέψεις. Παρουσιάζεται το έγγραφο αυτό στο Προεδρείο, κατόπιν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών πρόκειται επίσης ε, για την πολύ σημαντική φάση που ακολουθεί αυτή της ε, συζήτησης και συμφιλίωσης. Έγκριση από το Προεδρείο, από την Επιτροπή Προϋπολογισμού, είναι η φάση στην οποία βρισκόμαστε και κατόπιν στην Ολομέλεια. Όσον αφορά την προετοιμασία του προϋπολογισμού στην κάθε γενική διεύθυνση, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας όλες τις ε, κατευθυντήριες γραμμές που εσείς παρουσιάζετε. Πρέπει να βασιστούμε σε αρεαλιστική βάση. Να τηρήσουμε την δημοσιονομική πειθαρχία, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Η αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σαν μία από τις αρχές ε, της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού, εξαρτάται από τη δημοκρατική διαδικασία με την οποία λειτουργεί στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θέματα που αφορούν την προετοιμασία και την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Προσπαθούμε κάθε φορά να αναλύσουμε για κάθε γραμμή του προϋπολογισμού ποιες είναι οι δραστηριότητες που μπορεί να εγκαταληφθούν, ποια είναι τα προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί, ποιες είναι επαναλαμβανόμενες ε, παλιές δραστηριότητες και οι νέες δραστηριότητες οι οποίες θα πρέπει να εκτιμηθούν με πολύ συγκεκριμένα σημεία αναφοράς των αποφάσεων των πολιτικών για το 2020. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Πρόκειται για μια χρονιά μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Επανερχόμαστε στην κανονική λειτουργία του Κοινοβουλίου μετά από τη σύσταση της νέας Επιτροπής και κατόπιν κάποιες από τις αποζημιώσεις ε, του τέλους ε, μιας θητείας μπορεί να συνεχιστούν ακόμα και δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θητείας. Θέλω επίσης, αναφερόμενος σε αυτή τη διοικητική διαδικασία, να σας αναφέρω τα αποτελέσματα των ακροάσεων. Πριν την εξέταση της ε, έκθεσης του εισηγητή σας, που λαμβάνει χώρα αυτήν την εποχή, Βλέπετε τα ποσά που έχουν εγγραφεί πριν δηλαδή περάσουμε στη φάση της έγκρισης του προσχεδίου και υπάρχει δυνατότητα εδώ για μια σχετική μείωση των κονδυλίων. 25,3 εκατομμύρια ευρώ είναι η φετινή μείωση. 1,21% είναι το ποσοστό μείωσης των ε, συνολικά των κονδυλίων. Ας περάσουμε τώρα στις γενικές γραμμές αυτού του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 2020. Θα σας παρουσιάσω ποιες παράμετροι χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση αυτού του προϋπολογισμού, την πολυετή εξέλιξη του προϋπολογισμού σχέση με το τρίτο κεφάλαιο, η τα μεγάλα ποσά η κατανομή των ποσών μεταξύ των υποχρεωτικών δαπανών και των προσαρμόσιμων δαπανών, οι δαπάνες που αφορούν την πολυγλωσία, και εδώ θα αναφερθώ και στα θέματα που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Link και βεβαίως ε, οι πιστώσεις που ουσιαστικά διαχειρίζεται η κάθε Γενική Διεύθυνση ξεχωριστά. Όσον αφορά τις παραμέτρους, αυτό είναι καθοριστικό για να μπορέσει κάποιος να εκτιμήσει το σύνολο και τον όγκο των ε, κονδυλίων και των πιστώσεων. Θα πρέπει όλοι να έχουν την ίδια βάση, να καθοριστεί ένας ε, συγκεκριμένος αριθμός πολιτικών δραστηριοτήτων και να υπάρχει εναρμόνιση με των άλλων ε, θεσμικών οργάνων όσον αφορά τα ποσοστά και τους συντελεστές που θα εφαρμοστούν. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε εδώ, παραδείγματο χάρη για τον πληθωρισμό, ποσοστά τα οποία δεν είναι εναρμονισμένα. Η αύξηση, παραδείγματο χάρη των αποδοχών των συνεργατών του Κοινοβουλίου γίνεται βάσει μια συγκεκριμένης μεθόδου το ίδιο ισχύει και για τα συμβόλαια τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη. Λαμβάνουμε υπόψη μας την έδρα, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο για το κάθε συμβόλαιο, την κάθε σύμβαση. Εδώ σε αυτό το πίνακα σας υπενθυμίζουμε ακριβώς αυτούς τους συνταλλεστές. τον αριθμό των ε, δαπανών που αφορούν τις συνεδριάσεις, τις ολομέλειες, έκτακτες και τακτικές, καθώς και τις συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων τις εβδομάδες ε, όπου το Κοινοβούλιο συνεδριάζει εκτός Βρυξελών και Λουξεμβούργου. Πρόκειται για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν ε, τα έξοδα μετατόπισης των αντιπροσωπιών και των επιτροπών. Νομίζω ότι ο Γενικός Διευθυντής σας έχει παρουσιάσει πριν από λίγες μέρες αυτήν την, αυτό το πίνακα. Πρόκειται για τα τελευταία χρόνια. Για ποσά που φτάνουμε σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια 3,58% είναι το ποσοστό αύξησης όσον αφορά το κεφάλαιο 5. Οι διοικητικές δηλαδή δαπάνες έχει μειωθεί ενώ το 2019 με 2020 η αύξηση σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα φτάνει στο 4,34%. Το 2015 και επί 15 χρόνια το 20% αυτού του κεφαλαίου ήταν σταθερό αφιερωμένο στις δαπάνες αυτές. Όσον αφορά τα σημαντικά ποσά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 70% των δαπανών συγκεντρώνονται σε τρεις τομείς δαπανών. Το προσωπικό 35% μόνιμο προσωπικό, τα έξοδα των βουλευτών, 430 εκατομμύρια, και τρίτο κατηγορία δαπανών, οι ε, κτηριακές δαπάνες. Ένας άλλος πολύ σημαντικός τομέας αυτών των δαπανών, που είναι οι εξωτερικές γλωσσικές υπηρεσίες, 8%, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, 7%, οι πολιτικές ομάδες, τα ιδρύματα, 6% 128 εκατομμύρια. Δαπάνες που αφορούν την ενημέρωση, την πληροφορία 5% και κάποιες άλλες δευτερεύουσες διοικητικές δαπάνες, συνεδριάσεις ε, και άλλες δαπάνες προσωπικού. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το 70%, αυτό το ποσοστό των 70% που ουσιαστικά κατανέμεται μεταξύ των τριών αυτών τομέων με σχετικά σταθερό τρόπο όλα αυτά τα χρόνια. Παρουσιάζουμε μάλιστα και μια μικρή μείωση των μονίμων υπαλλήλων, τα 5% τα τελευταία χρόνια και μια μείωση όσον αφορά τις δαπάνες, ε, τις κτηριακές για τους περισσότερους τομείς. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση για σας είναι η αξιολόγηση των ε, υποχρεωτικών δαπανών καθώς και αυτών που ενδεχομένως ε, μπορούν να γίνουν αντικείμενα προσαρμογών. Οι υποχρεωτικές δαπάνες, μέλη του Κοινοβουλίου, προσωπικό, πολιτικές ομάδες, είναι το 73% του συνόλου των δαπανών. αυτές ε, προκαθορίζονται σε σχέση με πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Οι διοικητικές δαπάνες που αφορούν άλλα έξοδα, ενίκια, πολυετή, συντήρηση, καθαρισμός. Όλες αυτές οι συμβάσεις, οι πολυετής, για τις οποίες Υπάρχουν συντελεστές επανεκτίμηση και προσαρμογής οι οποίοι ορίζονται βάσει των συμβάσεων. 274 εκατομμύρια, 294 εκατομμύρια, συγγνώμη, είναι το 14% των ε, δαπανών, καθώς και οι λεγόμενες άλλες δαπάνες, οι οποίες δεν καθορίζονται βάσει κανονισμών, Βλέπετε όμως ότι περίπου το 85% των ε, δαπανών είναι ουσιαστικά υποχρεωτικές δαπάνες, επί των οποίων δεν υπάρχει περιθώριο ελιγμού και ευελιξία. Οι Γενικές Διευθύνσεις Link και Μετάφραση είναι εδώ σήμερα. Θα ακούσουμε λοιπόν μια γενική προσέγγιση για το θέμα της πολυγλωσσίας είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ε, θέμα αυτό γιατί βλέπετε ότι οι δαπάνες προσωπικού στις γενικές αυτές διευθύνσεις, link, φτάνουν τα 171 και 80 εκατομμύρια για τη μία και την άλλη. Κατόπιν έχουμε τους εξωτερικούς συνεργάτες, 8 εκατομμύρια για τις μεταφράσεις και 48 εκατομμύρια για τους ε, εξωτερικούς συνεργάτες στον τομέα της διερμηνίας, 439 εκατομμύρια συνολικό ποσό κόστος για την πολυγλωσία. Επί αυτών των άμεσων δαπανών θα πρέπει να προσθέσουμε και κάποιες έμεσες, 28 εκατομμύρια συνολικά η πολυγλωσία μας στοιχίζει 467 εκατομμύρια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για το 23% των δαπανών του Κοινοβουλίου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι κάτι το αμεληταίο. Εάν το συγκρίνουμε με το Εθνικό Κοινοβούλιο που δεν έχει αυτόν τον παράγοντα της πολυγλωσίας. 467 εκατομμύρια αφορούν την πολυγλωσία. Τέλος, η κατανομή των πιστώσεων στις διάφορες γενικές διευθύνσεις βλέπετε ότι σε σχέση με τα συνολικά ποσά, όπως σας παρουσίασα πριν από λίγα λεπτά, η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, ΠΕΡΣ, που είναι η πιο σημαντική διεύθυνση εδώ, ακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, ΦΙΝΣ, για τα έξοδα των ε, βουλευτών, κατόπιν ΙΝΛΟ, και οι υπόλοιπες διευθύνσεις ακολουθούν ανάλογα με την σημασία του τομέα τους. Αυτά όσον αφορά τις ε, γενικές κατευθυντήριες γραμμές για το 2020. Πολύ σύντομα θα σας κάνω μια παρουσίαση του τρίτου τμήματος που είναι τα τμήματα που διαχειρίζεται η δική μου γενική διεύθυνση, δηλαδή έξοδα που αφορούν ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου καθώς και τις πολιτικές ομάδες και τα ιδρύματα. Εδώ θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η συνδρομή στα μέλη του Κοινοβουλίου είναι η μεγαλύτερη δαπάνη πάνω από τις αμοιβέ των βουλευτών, πάνω από τα 70 δηλαδή εκατομμύρια και 74 εκατομμύρια για το 2020 τα έξοδα των μετακινήσεων. Θα πρέπει επίσης εδώ να σημειώσουμε ότι ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας και οι χώρες προέλευσης των ε, μελών του Κοινοβουλίου ουσιαστικά είναι ένα ποσό που αντιστοιχεί περίπου στις αποδοχές τους. Κατόπιν έχουμε τα γενικά έξοδα, 39 εκατομμύρια ευρώ, συντάξεις, αποζημιώσεις που θα είναι πιο υψηλές το 2019 γιατί κάποιοι όταν αλλάξει το κοινοβούλιο μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές θα αποζημιωθούν και η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ μειωμένο αυτό το ποσό, 13 εκατομμύρια. Τέλος, η κατανομή των ε, δαπανών που αφορούν τα πολιτικά, τις πολιτικές ομάδες και τα ιδρύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άμεσες πιστώσεις στα στις πολιτικές ομάδες, 65 εκατομμύρια ευρώ, η χρηματοδότηση των ε, ευρωπαϊκών πολιτικών ε, ομάδων και των ιδρυμάτων αντιστοιχεί το ποσό των 63 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε στο κόστος ε, των πολιτικών ομάδων το προσωπικό των πολιτικών ομάδων που καλύπτεται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό 136 εκατομμύρια ευρώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κλεφή. Και τώρα, οι σκιώδεις έχουν μήπως ερωτήσεις να απευθύνουν. Ο κ. Μανκά, ο εισηγητής. Αν έχετε ερωτήσεις σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Λεφή, για την πολύ καλή παρουσίαση ε, των στοιχείων. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά που κάνει η Γενική του Διεύθυνση. Τα ερωτήματα θα απευθυνθούν περισσότερο προς τη συνάδελφό σας, την κυρία Λίνς, γιατί και πάνε τα περισσότερα κονδύλια. Ένα σχόλιο για όλες τις γενικές διευθύνσεις όμως είναι αυτό που θα αναφέρω τώρα. Ε, πρέπει, ξέρετε, μια φορά κάθε, μετά από κάποια χρόνια να ρίχνουμε μια καλή ματιά για να δούμε τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, πώς πάει. Από καιρού εις καιρών είναι καλό να εντοπίζουμε κάποια σημεία προσβελτίωση βελτίωση της συνεργασίας, όπως πληροφορική, ασφάλεια, μετάφραση, μεταφραστικές υπηρεσίες, υπηρεσία οδηγών και κάποιε άλλε υπηρεσίε. Είναι μια ερώτηση. Και στο Προεδρείο έθεσα το ερώτημα στο Γενικό Γραμματέα και είπε ότι υπάρχουν κάποια αποθέματα, κάποια, ε, ε, κάποια στον τομέα των οδηγών μπορούμε να έχουμε κοινή χρήση του προσωπικού ε, και με αυτόν τον τρόπο να πετύχουμε κάποιες οικονομίες. Λοιπόν, αυτή είναι η ερώτηση προ του γενικού διευθυντέ. Υπάρχει τη δυνατότητα συνεργασία κοινή χρήση του προσωπικού των θεσμικών οργάνων. Συζητήσαμε το θέμα με του Κιώδη και ένα θέμα διεφάνει. Είδαμε ότι στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε και την επεξήγηση ψήφων, όπου οι βουλευτές επεξηγούν την ψήφο τους και χρησιμοποιούν το χρόνο για να προβληθούν, να παρουσιαστούν, μιλούν τη γλώσσα, στη γλώσσα τους, δεν υποβάλλονται ερωτήσεις. Εάν υπολογίσουμε αυτό, πόσο κοστίζει, η επεξήγηση ψήφου, και εκ... ήταν εκεί και ο Ρούμπικ και εκπρόσωποι της Άλντε όταν το συζητήσαμε αυτό και είπαμε ότι ίσως μπορούμε να εγκαταλείψουμε την επεξήγηση ψήφου διότι οι ευρωβουλευτές μπορούν να εξηγήσουν την ψήφο τους με άλλους τρόπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο μας κοστίζει η επεξήγηση ψήφου. Έχω και κάποια δική μου προσωπική ε, πρόταση, αλλά έχει τα όρια της. Παραδείγματο χάρη, αν δεν υπήρχε διερμηνία, Φερρυπίν, τι θα συνέβαινε. Ο πρόεδρος ίσως της Ολομέλειας δεν θα κατανοούσε τι λένε οι ευρωβουλευτές και τι εξηγούν, ποια είναι η εξήγηση που δίνουν. Όμως θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε και στις οικονομίες. Ε, και θα θέσω και άλλες ερωτήσεις. Πριν από αυτό όμως, να πω κάτι άλλο. Πριν από κάποια χρόνια, είχαμε πολλές γραπτές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτριετίας Φερρυπίν και λάβαμε κάποια μέτρα και μειώσαμε τον αριθμό των ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τις μειώσαμε κατά 70% σε τρία χρόνια. 9.000 ερωτήσεις ή λιγότερες έχουμε τώρα. Άρα 6,3 εκατομμύρια ευρώ. 40% είναι η οικονομία του Κοινοβουλίου και τα υπόλοιπα είναι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτοί που επεξεργάζονται τις ερωτήσεις, οι δεκάδες άνθρωποι χρειάζονται για να σε επεξεργαστούν. Μειώθηκε από τη μείωση του αριθμού των ερωτήσεων. Είχαμε κάποια μείωση προσωπικού. Κάναμε κάποιε οικονομίε όσον αφορά το προσωπικό. Αν δεν θέλουμε να βασίζουμε σε κάποιου δείκτε αποκλειστικά τον προπολογισμό, εντάξει, μπορούμε να κινηθούμε μόνο βάσει στοιχείων. Αλλά, ερώτηση μπορούμε να κάνουμε κάποιες οικονομίες. Εάν υπάρξει κάλυψη από κάποια άλλα ε, σημεία του προπολογισμού. Ευχαριστούμε. πολύ κύριε Μάνκα. Συγγνώμη όμως, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσω εδώ κάτι. Αρχικά είχαμε μια σειρά. Πρώτα να ακούσουμε δηλαδή και τις πέντε γενικές διευθύνσεις, τους εκπροσώπους αυτών, να μας παρουσιάσουν τα θέματά τους καθεμία και να επακολουθήσουν οι ερωτήσεις για την κάθε γάμα δέλτα μετά από την παρέμβαση κάθε γάμα δέλτα. Τώρα δεν ξέρω, επειδή είστε εισηγητής και είστε αυτός που διατάζει, αν δεν σας δημιουργεί αυτό πρόβλημα, να ακούσουμε πρώτα και τις πέντε γαμαδέλα και μετά να ακούσουμε τις ερωτήσεις, δηλαδή να ξαναγυρίσουμε στην αρχική ημερήσια διάταξη και σειρά. Τούτους συναδέλφους και πρώτα τους κοιόδες ερωτώ λοιπόν, εάν θέλουν να ρωτήσουν κάτι τη γάμα δέλτα οικονομικά, finance. Ευχαριστώ πολύ, πολύ γρήγορα. Το είχα ρωτήσει και την προηγούμενη φορά που μας παρουσίασε τον προπολογισμό Γενικός Γραμματέα. Δεν έχουμε όμω πολύ χρόνο, μάλλον τότε δεν είχαμε πολύ χρόνο και έφυγε και δεν άκουσα να δεν υπήρξε απάντηση. Προβλέπεται ο πληθωρισμό ε, για το 2020 στις διαφορες έδρε έδρες 1,6-1,8. Εκεί κυμαίνεται. Και για την αναπροσαρμογή των μισθών και των δαπανών για τους βουλευτές χρησιμοποιείται το 1,8%. Όμως, ε, αν κατάλαβα καλά την προηγούμενη φορά και θέλω το βλέπω και στο πλαίσιο στους πίνακες, ότι για την αναπροσαρμογή ε, των δαπανών του προσωπικού χρησιμοποιείται το 2,5%. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά όταν έχουμε εκτιμήσεις που μιλάνε για ένα επίπεδο πληθωρισμού μεταξύ 1,6 και 1,8 <coughs> Ουσιαστικά πρέπει να φασιζόμαστε ε, σε αυτό και είναι σημαντικά και τα δεκαδικά ψηφία για τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν γιατί έχουμε αυτή τη διαφορά. Άλλες ερωτήσεις. Αν όχι, εγώ έχω μια ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος, πάρα πολύ σύντομα. Θα ήθελα να μας δώσετε κάποια στοιχεία για την πρόταση περί διατήρησης ε, των συμβασιούχων, ακόμη και μετά το τέλος ε, της ε, εκλογικής περίοδου που θα προσληφθούν για τις εκλογές και θα πάνε ε, μετά σε θέση AST για τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι 51 άτομα και 51 θέσεις δηλαδή. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, μετά τα, τις θέσεις αυτές μάλλον, μετά από το Ιούνιο πού θα πάνε και με τι καθήκοντα. Και ίσως το σημαντικότερο, αυτό συνεπάγεται και αύξηση στο οργανόγραμμα Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σε το πρώτο ερώτημα που αφορά τον πληθωρισμό. Πράγματι, πρέπει να εφαρμόσουμε για τις διάφορες δαπάνες ε, το ποσοστό πληθωρισμού που προβλέπει ο ισιών κανονισμός. Αυτό τι σημαίνει για τις αποδοχές ε, των υπαλλήλων και των βουλευτών προβλέπεται στο καταστατικό ε, για τη δημόσια διοίκηση ο υπολογισμός που εγκρίθηκε από κοινού από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο κατά την τελευταία αναθεώρηση του καθεστώτος δημόσιας διοίκησης και σε ένα καλό αλλά αν θέλετε, βλέπουμε πώ εξελίσσεται η αγοραστική δύναμη των υπαλλήλων σε ορισμένε χώρε, των δημόσιων υπαλλήλων σε ορισμένε χώρε. Αυτή η μέθοδο είναι και επικυρωμένη επιστημονικό αλλά και πολιτικό, εφόσον έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος, του καταστατικού ε, των βουλευτών, οι οποίοι αμείβονται με ένα ποσοστό του μισθού των δικαστών και υπάρχει αυτό το ποσοστό αναπροσαρμογής που ορίζεται κάθε Δεκέμβρη και αρχίζει να ισχύει από τον Ιούλιο κάθε τρέχοντος έτους. Άρα για τον προπλησμό του 2020 προβλέπει η Κομισιόν αυτή τη στιγμή ε, ότι θα είναι 2,5 αυτό το ποσοστό και όλα τα θεσμικά όργανα έχουν υπολογίσει αυτό το ποσοστό. Αν αλλάξει, που κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, στη διάρκεια των συνδιαλλαγών ε, για το σχέδιο, ή μάλλον όταν εγκριθεί το σχέδιο περιπολισμού τον Οκτώβριο, εκεί μπορεί να γίνουν προσαρμογέ. με βάση το τελευταίο γνωστό νούμερο. Στο δεύτερο το 1,8%. Αυτό το νούμερο απορρέει από κάποια μέτρα εφαρμογή του καταστατικού που λένε ότι όλες οι λοιπές ε, δαπάνες για τους βουλευτές, δηλαδή χιλιομετρική αποστάση τα οδηπαρικά δηλαδή, αποζημίωση γενικών ε, εξόδων ε, και η αποζημίωση για τη διάρκεια κτλ. βασίζεται σε αυτά τα οποία ίσχυαν τον Οκτώβριο νήμιον 1 και νη έτους. Τι προβλέπουμε λοιπόν για τον φθινόπωρο του 18 από την Κομισιόν. Ε, προβλέπεται 1,8% και αυτό θα ισχύει για το 2020. Βέβαια, εμείς θα πάρουμε ε, για την εκτέλεση το το δημοσιευθένα ποσοστό. Το Νοέμβριο θα ξέρουμε ποιος ήταν, ποιο ήταν το ποσοστό πληθωρισμού από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι τον Οκτώβριο του 2019. Και αυτό θα εφαρμόσουμε. Υπάρχει απόφαση του Προεδρείου που ε, λαμβάνεται το Δεκέμβριο και αυτόν το νέο ποσοστό το υπολογίζουμε για τις αλληλεπές δαπάνες των βουλευτών σε ό,τι αφορά τους εμβασιούχους οι οποίοι ε, θα είναι για τα γραφεία του Κοινοβουλίου στις διάφορες χώρες. Είναι 51 όπως είπατε και έχουν μια συγκεκριμένη αποστολή σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας για τις ευρωεκλογέ, να έχουν πιο άμεσες επαφές με την κοινωνία των πολιτών δηλαδή αυτά τα άτομα. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας επικοινωνία η οποία αξιολόγησε τα πρώτα αποτελέσματα των υπαλλήλων αυτών που έχουν αποσπαστεί ήδη από τον Ιούνιο του 2018. Ήταν τόσο ικανοποιητική η πρωτοβουλία και οι πρωτοβουλίες γενικά που ανέλαβαν αυτοί οι υπάλληλοι που έχει ζητηθεί ήδη να παραμείνουν και μετά τις εκλογές εκεί για να συνεχίσουν τις επαφές με τα κοινωνικά δίκτυα, την κοινωνία των πολιτών εν γέννη, για τις θέσεις ΑΕΣΤΕ. Θα πηγαίνουν στα γραφεία πληροφοριών ε, οι θέσεις αυτές που απελευθερώνονται. Κατά το ίμιση θα επανέλθουν στην Digicom και κατά το ίμιση σε άλλες υπηρεσίες οι θέσεις αυτές θα απελευθερώνονται. Thank Σας ευχαριστώ. Επόμενη Γενική Διεύθυνση, Γενική Διεύθυνση Ίνλο. Κύριε Λίντους, έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να παρουσιάσω κάποιες λεπτομέρειες μετά την παρουσία που έκανε Γενικό Διευθυντή στα στοιχεία. Να παρουσιάσω το τμήμα του προπολογισμού, το δικό μας, μετά την έξοχη παρουσίαση του Didier η DG Inlo είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακούσατε κάτι πρόσφατα και θέλω να το επενθυμίσω. Ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις από το Προεδρείο τον Απρίλιο του 2018. Ήρθε εδώ Γενικός Γραμματέας στην Επιτροπή Προπολογισμών και παρουσίασε τον Ιούλιο του 2018 αυτά τα στοιχεία. Είναι η νέα στρατηγική για τα κτίρια που παρουσίασε. Με τίτλο πέρα μετά το 2019. Ο προπολογισμό του 2020 είναι ο πρώτος προπολογισμό που εφαρμόζει αυτές τις αρχές που έχουν περιγραφεί στη νέα στρατηγική. Να υπενθυμίσω τις αρχές τέσσερις τον αριθμό. Να προσαρμοστούν οι εγκαταστάσεις στην εξέλιξη των συνεδριάσεων και να προσαρμοστούν οι αίθουσες ε, ανάλογα με τους θεσμοθετηθέντες τριμερείς διαλόγους, να κινηθούν πιο κοντά στους πολίτες. Η ευρωπαϊκή εμπειρία ε, μέσω των γραφείων συνδέσμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διάφορε να το πετύχουμε αυτό. Τρίτον, να συνεχιστεί η βελτίωση της ασφάλειας σε στενή συνεργασία τη Γενική Διευθύνσεως ΣΕΙΦ, αυτό αφορά τα κτίρια του Κοινοβουλίου, και να κλείσουμε κάποια κενά που υπάρχουν στις διασυνδέσεις των κεντρικών ε, κτηρίων, κυρίως στις Βρυξέλλες. Όπως είδατε ή ακούσατε από την παρουσίαση του κυρίου Κρεσί, κάποια ποσά που διατίθεται για το Κοινοβούλιο αφορούν μισθολογικά έξοδα και οι δαπάνε είναι αρκετά γραμμικέ. Και εκεί ο, η κατάρτιση του προπολογισμού είναι αρκετά απλή. Η γενική διεύθυνση law είναι κάπω διαφορετική. Διότι τα δικά μας κονδύλια δεν είναι γραμμικά. Γιατί. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιούμε τα χρήματα του υπολογισμού μέσω ε, διαγωνισμών. Έχουμε πάνω από 600 ε, συμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί διαφόρων μεγεθών για διάφορες υπηρεσίες που ποικίλουν από catering μέχρι υπηρεσία αυτοκινήτων, κτηριακά προγράμματα, έργα συντήρησης και βέβαια η τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός των κτηρίων. Εν να πω, διότι εδώ θα είναι τελευταία παρουσίασή μου εδώ, σε αυτή τη θητεία, να σας πω κάποια πράγματα που κάναμε στον φατοπυρπολογισμό μαζί με το Προεδρείο. Σε κάποιους τομείς κάναμε σημαντικές οικονομίες, χάρη στις συμβουλές σας. Μειώσαμε τα κονδύλια. Ένα παράδειγμα. Catering. Το 2014 ήμασταν κοντά στα 5 εκατομμυρία χορηγουμένων υπηρεσιών catering. Τώρα είμαστε 0,8 εκατομμύρια. 800.000 ευρώ. Δεν υπάρχει επιχορήγηση συμβάσεων πλέον. Αλλά έχει κάποιες ευθύνες στο Κοινοβούλιο. Για φιλανθρωπικές δωρεές κλπ. Για άλλα στοιχεία. Αυξήθηκαν τα κονδύλια εσωτερικεύση των υπηρεσίες αυτοκινήτων. Φερρυπίν. Όταν ήταν συγγητής ο κ. Ρούμπικ, το εξετάσαμε αυτό, αυξήθηκε ο προπολογισμό κατά 3-4 εκατομμύρια, αν θυμάμαι σωστά. Με σαφή μείωση διαμαρτυριών από τους πελάτες όμως έχει βελτιωθεί κατά πολύ η παροχή των υπηρεσιών, με άλλα λόγια. Το 2020, ο προπολογισμό του 2020, τι ζητάμε. 238,36 εκατομμύρια ευρώ. εξηγούνται κάποιες αυξήσεις λόγω της ιδιαιτερότητας του έρτους. για την ολοκλήρωση του κτηρίου ΚΑΝΤ στο Λουξεμβούργο όπου γίνεται η μετακόμιση υπάρχουν θέματα για μίσθωση του κτηρίου και, μετα... και τα έξοδα μετακόμιση από το παλιό στο νέο κτίριο. Άλλη αύξηση οφείλεται στη νέα πολιτική για την εμπειρία Ευρώπα. Προτείνουμε πέντε νέα γραφεία συνδέσμους στην περιοχή, στις ειδικέ περιοχές για τις επαφές με τους πολίτες. Πρέπει να γίνει προετοιμασία για ανακαίνιση του κτηρίου ΣΠΑΚ Πρέπει να ολοκληρωθεί και το επενδυτικό σχέδιο για την ασφάλεια και το κονδύλι για τα έπιπλα και τον εξοπλισμό. Στο τέλος θα δώσω περισσότερες εξηγήσει. Να σας πω τι γίνεται με τα γραφεία των μελών. Για το CAD. Conrad το κτίριο Conrad Adenauer. Η Ανατολική Πτέρυγα έχει ολοκληρωθεί που είναι η μεγαλύτερη και έχει τα περισσότερα γραφεία στο Λουξεμβούργο. Το Δεκέμβριο φέτος θα τελειώσουν οι εργασίες. Και έχουμε διάφορες δαπάνες σχετικές. Πρώτα απ' όλα δαπάνες με, να κενωθεί το κτίριο, τα, τα, μετά τα έπιπλα, μετα, μάλλον μαλλον έπιπλα, ενέργεια, γιατί έχουμε και την μίσθωση των δύο πύργων που έχουμε μισθωμένους τους πύργους από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου. Με τα χαράς, λέγω και συγχαίρω τους συναδέλφους για το εξή. Η αρχή του προπολογισμού το 2009 έδωσε 432 εκατομμύρια, καθόρισε 432 εκατομμύρια για τα έργα οικοδόμησης, οικοδομών και είμαστε κατά 20 ε, εκατομμύρια κάτω από αυτό το όριο, παρά τα προβλήματα. Υπάρχει και ένα κόστος ε, για λόγους αρχιτεκτονικών σχεδίων κλπ. Και, και ξεπεράσουμε αυτό το όριο. Αλλά έχει συγκρατηθεί το κόστος για τις οικοδομές. Αυτή ήταν πάντα η προσέγγιση που ακολούθησε και το Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Αν ξεπεράσουμε το όριο, θα έπρεπε να γίνουν και διάφορες προσαρμογές. Προετοιμασία για το Paul Henry Να Επενθυμίσω κάποια πράγματα. Ιούλιος 2018. Το Προεδρείο έλαβε απόφαση. Εκλήθη ο Γενικός Γραμματέας και η Γενική Διεύθυνση ΙΛΟ να ξεκινήσουν διαγωνισμό αρχιτεκτονικό για την ανακαίνιση του κτηρίου. Δύο επιλογές υπήρχαν μία εις βάθος ανακαίνιση, μία ριζική ανακαίνιση και μία εκ νέου οικοδόμηση του κτίριου. Τελική απόφαση μετά το διαγωνισμό. Μάλλον προετοιμάζεται ο διαγωνισμός. Ενδιαφέρονται διάφορες γενικές διευθύνσεις. Η πρόταση θα παρουσιαστεί το 2019, τέλος 2019, αρχές του 2020 θα υποβληθεί η πρόταση στο Προεδρείο προς απόφαση. Θα διαλέξει α ή β, ανακαίνιση ή ανοικοδόμηση. Ποια είναι τα προπαρασκευαστικά στάδια και οι σχετικές δαπάνες. Πρώτα απ' όλα, χρειάζονται τεχνικές μελέτες. 2,1 εκατομμύρια υπολογίζεται θα κοστίσουν. Μετά έχουμε το μετρήσει, θέλουμε επιστοποίηση για τα έργα σχέση με το περιβάλλον 1,2 εκατομμύρια περιβαλλοντικές αποδόσεις και 8,8 εκατομμύρια άλλα, άλλα συναφή έργα. Κάποιες λειτουργίες αυτού του κτηρίου θα μετακινηθούν. Όταν ξεκινήσουν τα έργα, θέλουμε, βλέπετε, να έχουμε έθεση συνεδριάσεων για το Προεδρείο και για τους κοσμήτορες και για τη διάσκεψη των Προέδρων. Πρέπει να γίνονται κάποιες λειτουργίες. Τεχνική αίθουσα για την DG Links, για τις τεχνικές υπηρεσίες, ο βασικός κόμβος, ε, είσοδο για το πρωτόκολλο, υπηρεσίες για τον τύπο και για τα ΜΜΕ, και είσοδο για τα ΜΜΕ. Το γραφείο του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα πρέπει να αντικατασταθούν, να μεταφερθούν. Οπτικοακουστικά έργα και τεχνικές λειτουργίες θα μετακινηθούν σε άλλα κτίρια. Και αυτό κοστίζει. Ασφάλεια. Θα είμαι σύντομη γιατί ξεπέρασα το χρονικό μόριο. Ασφάλεια. Θα πρέπει να έτοιμο το κτίριο ε, το 2020 στο Στρασβούργο για το Europe Experience. Πέντε νέα εγκαταστάσεις το 2020. Λουξεμβούργο και Βαρσοβία, κόστος 2 εκατομμύρια κάθε εγκατάσταση. Δουβλίνο, Χόλμη και Πράγα, 1,2 εκατομμύρια κάθε κτηριάκι για, τις, για την παρουσίαση του ευρωπαϊκού εγχειρήματο Europe Experience. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό για σας. Έπιπλα. Εξοπλισμός. Δύο παράλληλες πορείες ακολουθούμε εκεί. Το 2014 πήγατε στα γραφεία σας και υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες. 2.300 διαμαρτυρίες έφτασαν στην DG Inlo για αλλαγή επίπλων για γραφείο το οποίο δεν ικανοποιούσε το προσωπικό ή τον Ευρωβουλευτή. Έγινε μεγάλη προσπάθεια. Γίνονται έργα συντήρησης. Κατασκευάζουμε αίθουσε συνεδριάσεις. χώρους συνάντησης στους διαδρόμους, αλλάζουμε τα χαλιά, βάφουμε τους διαδρόμους και τα γραφεία για να είναι έτοιμα τα γραφεία μετά τις εκλογές. Το πιο σημαντικό, τα έπιπλα των μελών που είναι παλιά, πάνω από 20 ετών, δηλαδή έχει πλέον παραγραφεί το χρέος τους, θα, θα την κατασταθούν μέσω μίσθωσης. Ύψος 3,6 εκατομμύρια το χρόνο το κόστος μίσθωσης. Χωρίς να αναφέρω λεπτομέρειες. Έχω υπογράψει την ανάθεση της μίστος αλλά έχουμε 10, μέρες περίοδο αναμονής. Δεν ξέρω πόσο θα κατέβουμε από το ποσό, το ποσό όμως θα συρρυκνωθεί αρκετά από το προβλεπόμενο. Δεκαετής θα είναι η μίστοση και μπορεί να παραταθεί και να γίνει δεκαπενταετής Θα είναι πιο φιλικά τα έπιπλα προς το χρήστη, καλύτερα από πλευράς περιβαλλοντικής, εργονομικής και θα καλύπτουν τις ανάγκες των μελών και του προσωπικού. Για πρώτη φορά χρησιμοποίησαμε διαφορετική διαδικασία ανάθεσης και διαγωνισμού. Ε, έλαβε χώρα διάλογος, απέδωσε καλά αποτελέσματα, ήταν μεγαλύτερος ανταγωνισμός που κατέληξε καλύτερα αποτελέσματα. Οι άλλες δαπάνες για τα έπιπλα σχετίζονται για την μετακόμιση προς το ΚΑΔ και ένα νεοκτήριο προφανώς πρέπει να επιπλωθεί. 4 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα παραπάνω χρειάστηκα. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ για την προσοχή σα και είμαι ανοιχτή προ υποβολή ερωτήσεων. Um, ευχαριστώ κύριε Λίνου. Και τώρα θα κάνω το εξή. Θα ζητήσω τον εισηγητή μετά από κάθε γενική διεύθυνση αν έχει συγκεκριμένη ερώτηση να υποβάλει προς συγκεκριμένη γενική διεύθυνση. Κύριε Μάνκα, έχετε ερώτηση. Ano, Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ απαιτητική αυτή η Γενική Διεύθυνση. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Λίνος για την εξαντλητική της παρουσίαση. Και πολύ πλήρη. Η πρώτη μου ερώτηση είναι εξής. Το Europe Experience θα οργανωθεί στην Πράγα, στη Στοκόλμη, στο Λουξεμβούργο και στη Βαρσοβία. Το Λουξεμβούργο είναι μια χώρα με 590.000 κατοίκους, μια μικρή χώρα, τέσσερις φορές πιο μικρή από τη Στοκόλμη, παραδείγματος χάρη. Βλέπουμε όμως ότι εδώ αναφερόμαστε σε ένα ποσό 1,4 εκατομμύρια. Μήπως πρέπει να οργανωθεί κάτι λίγο πιο μικρό στο Λουξεμβούργο. Γιατί να προβλέψουμε ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα πάει να επισκεφτεί το Λουξεμβούργο για να, δει το visit, για να επισκεφτεί το Europe Experience. Έχω και μια άλλη ερώτηση. Θα δοκιμάσουμε αυτά τα μοντέλα. Θα υπάρχουν και πειραματικά σχόλια και πιστεύω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι το θετικό πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ξέρουμε όμως που θα εγκατασταθούν οι πρώτες πιλωτικές αυτές εγκαταστάσεις. Και σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιωθεί η κατάσταση πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Όσον αφορά τα έπιπλα για το 2019, φέτος θα έρθουν νέα μέλη, νέοι βοηθοί. Πώς μπορούμε εδώ να εξοικονομήσουμε 6-8 εκατομμύρια βλέπω να έχετε προβλέψει. Είπατε ότι μπορεί το ποσό αυτό να μειωθεί. Χαίρομαι που το ακούω. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξουν ε, εξοικονομήσεις σε αυτή την κατηγορία. Το κτίριο PHS, αυτό το ρώτησαν και οι σκιώδεις ηγητές, τα 11 εκατομμύρια που προβλέπονται. Αναρωτιέμαι αν θα χρειαστούν, διότι από ό,τι καταλαβαίνω θα πρέπει να διάσει το κτίριο, όποια και να είναι η εναλλακτική λύση που θα επιλεγεί. Ε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρούμπικ, που είναι ο σκιώδης. Θα πρέπει να περιορίσουμε όμως ε, τις ερωτήσεις, γιατί αλλιώς θα ξεπράσουμε το χρόνο που έχουμε προβλέψει. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές από τις ερωτήσεις που θα ήθελα να κάνω προς αυτή τη νέα διεύθυνση, η οποία πραγματικά θεωρώ ότι πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι το θέμα των ταξιδιών, το θέμα των εγγράφων, των δικαιολογητικών που πραγματικά μέχρι τώρα μας απασχόλησε και ήταν ένας μεγάλος όγκος εργασίας. Σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχει μια αρχιοθέτηση η οποία γίνεται με αυτόματο τρόπο πολύ πιο απλό, πολύ πιο σύντομο. Θα ήθελα λοιπόν να σας συγχαρώ γιατί κατάλαβα ότι και η πρώτη φάση του λανσαρίσματος πήγε πολύ καλά. Έχουμε πλήρη ενημέρωση και για τις ε, μετακινήσεις με τρένο και με το αεροπλάνο αυτό που είναι το πιο σημαντικό για μας είναι να έχουμε μία συγκεκριμένη εικόνα όλων των μηνυμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται. Μπορείτε να μας πείτε εσείς ποια είναι η δική σας εμπειρία. Πολύ σύντομα, παρακαλώ, 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το Europe Experience στο Δουβλίνο, Θα είμαστε έτοιμοι μέχρι το 2020. Υπάρχουν δύο εκατομμύρια τα οποία έχουν ε, αφιερωθεί. Θα παραμείνει το ποσό αυτό ή πρέπει να το μεταφέρουμε στον επόμενο χρόνο. Κυρία Λίνος. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ γιατί ίσως μπορώ με αυτόν τον τρόπο να αποσαφηνίσω κάποια σημεία το Europe Experience. Θα ξεκινήσω με αυτό του Δουβλίνου. Ήμασταν σε επίσημη επίσκεψη με τον αντιπρόεδρο, τον ε, υπεύθυνο για τα κτίρια και τον ε, αρμόδιο ε, αντιπρόεδρο τον Ιρλανδό Δεν θέλω τώρα να εκφράσω ενθουσιασμό, θα το κάνω παρόλα αυτά. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό κτίριο, το οποίο είναι ακριβό, πιο ακριβό από αυτό που καταβάλουμε σήμερα βάσει της συμφωνίας που έχουμε με την Επιτροπή θα πρέπει να εγκατασταθεί και το Europa Experience. Είμαστε πραγματικά πολύ ευτυχείς με την επιλογή αυτή και στην επόμενη συνάντησή μας, 13 ε, Μαρτίου του 2019, στη συνεδρίαση με αντικείμενο την κτηριακή πολιτική, θα παρουσιάσουμε το ε, κτίριο αυτό. Ελπίζω να είμαστε εντάξει όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τα χρήματα αυτά σίγουρα θα τα χρειαστούμε. Για το Λουξεμβούργο υπάρχουν δύο λόγοι που έχουμε προτείνει αυτήν την μεγαλύτερη, αν θέλετε, δυνατότητα εγκατάστασης. Στο παρόν κτίριο, ουσιαστικά στο οποίο θα εγκατασταθεί το Europe Facility, δεν είναι κάτι που θα προκαλέσει επιπλέον έξοδο. Και όσον αφορά το Λουξεμβούργο, το Λουξεμβούργο είναι μια πολύ ειδική περίπτωση χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει στο Λουξεμβούργο, προκαλεί επισκέψεις και ενδιαφέρον, δραστηριότητες με τις αρχές του Λουξεμβούργου οι οποίοι πραγματικά στο χώρο του Κίρσμπεργκ έχουν δραστηριοποιηθεί σε πολλά επίπεδα. Τώρα, το άλλο θέμα που δείξατε και το οποίο αφορά τις μετακινήσεις των ε, βουλευτών. Κύριε Μάνκα, θα την μεταφέρω στους ε, συναδέλφους από την Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας. Δεν είναι δική μας αρμεδιότητα. Ξέρω ότι κινείται πάντως το θέμα. Το θέμα τώρα των ε, επίπλων και οι πιθανές εξοικονομήσεις. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θέλουμε να υπάρξουν σημαντικές ε, εξοικονομήσεις. Όχι οριακές και βεβαίως όλοι αυτοί που πρέπει να εγκατασταθούν στο Λουξεμβούργο θα το κάνουν στο νέο κτίριο, με νέα κτίρια και με νέα έπιπλα. Σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε για το PHS. Όντως, πρέπει να γίνουν ε, κάποιες εργασίες εδώ σε αυτό το κτίριο και γι' αυτό και χρειάζεται και αυτή η προετοιμασία. Κύριε Ρούμπιχ, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για το Luling Lounge. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τα μέλη, για τους συνεργάτες. Όλα αυτά βεβαίως περιέχονται στις προτάσεις μας. Δεν θέλω να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά κάπως έτσι αλλάζουμε τα κτίρια μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις υπηρεσίες. Είναι πολύ καλό το σχόλιο σας επίσης ε, όσον αφορά τα νέα κτίρια και τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Τους οδηγούς υπάρχουν ε, συζητήσεις μεταξύ των δύο γενικών διευθύνσεων και ελπίζω τα μέλη να έχουν λίγο πιο απλές εφαρμογές για το θέμα των οδηγών, αλλά χρειάζεται και η προστασία των δεδομένων και θα πρέπει η εφαρμογή που χρησιμοποιούν τα μέλη του Κοινοβουλίου να είναι αξιόπιστη, ασφαλής και θα το εξετάσουμε και αυτό το θέμα τους επόμενους μήνες. Ευχαριστούμε την κυρία Κλίνους και προχωρούμε στην επόμενη Γενική Διεύθυνση για να μην βγούμε εκτός χρόνου. Γάμα Δέλτα Σέιφ, Έλιο Καρότσα, ο Γενικός Διευθυντής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να σας παρουσιάσω τον προπολισμό της Χαμάτλητα Safe και ταυτόχρονα να σας παρουσιάσω και τη γενική μας διεύθυνση. Όπως είπε και ο κύριος Κλετή, σε σχέση και με τον προπολισμό της ΓΑΜΑΤΛΤΑ ήλιο θα δείτε ότι η ΓΑΜΑΤΛΤΑ Safe δεν έχει ένα μεγάλο προπολογισμό, όμως σε σχέση με τα αριθμητικά στοιχεία και για τη ΓΔ δεν πρέπει να υποτιμούμε το γεγονός ότι ένα σημαντικό τμήμα του ε, προπολογισμού αφορά ε, τη διαχείριση της ΓΔ ΠΕΡΣ, μέσω της οποίας πληρώνονται οι υπάλληλοι ε, φύλακες, που πλέον είναι μια εσωτερική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Η ΓΔ ΣΕΙΦ ε, συρρυκνούνται Άλλες ε, θέσεις αυξάνονται, άλλες μειώνονται. Αυξάνονται οι θέσεις που σχετίζονται με την ε, πυρασφάλεια σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο και για τη Γενική Γραμματεία του, του Ξεμβούργου. Πάλι πυρασφάλεια και αυτές οι αυξήσεις αιτιολογούνται από την αύξηση του δίκτυ που το 19 και το 20 έχει έχει υπολογιστεί ε, και οι άλλες αυξήσεις έχουν να κάνουν με την επέκταση της περιμέτρου και αφορούν το Στρασβούργο. Διότι με τη νέα πολιτική να είναι ανοιχτά τα κτίρια του Στρασβούργου εκτός περιόδων Λομέλειας, οπότε να υπάρχει δυνατότητα εκεί να παραχωρούνται κάποιες αίθουσε σε διάφορες συνεδριάσεις μπορεί να έχουμε μια πιο μαζική παρουσία και χρειάζεται λοιπόν πυρασφάλεια, πυροσβεστική και στις Βρυξέλλες έχουμε μια ελαφριά αύξηση λόγω της αύξησης του δίκτυου, δηλαδή τη μαριθμική αναπροσαρμογή αλλά και έχουμε μεγαλύτερη περίμετρο γιατί ο παιδικός σταθμός ε, των Βρυξελών επεκτάθηκε. Επίσης, και θέλω να σας ευχαριστήσω που το έχετε υπογραμμίσει, το Λουξεμβούργο σε σχέση με Στρασβού και Βρυξέλλες έχει ένα πολύ μεγαλύτερο προπολογισμό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμη προχωρήσει σε στερική ανάθεση των υπηρεσιών. Δεν το ξεχάσαμε, απλά περιμέναμε ε, να υπάρξει μια μεταφορά, ε, να γίνει δηλαδή μετακόμιση στο ΚΑΝΤ, στο καινούριο κτίριο, για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες ε, οικονομίες και ένα πολύ μεγαλύτερο εξορθολογισμό των δαπανών σε σχέση με την κατάσταση ως ισχύει σήμερα στο Λουξεμβούργο. Αν δηλαδή είχε γίνει αυτή η εσωτερήκευση, αν μπορώ να το πω έτσι, με βάση τα υφιστάμενα σήμερα κτίρια, θα χρειαζόταν να είχαμε δαπανίσει το διπλάσιο από αυτό που θα δαπανίσουμε μετά το 2021, οπότε δηλαδή οι υπηρεσίες μας θα έχουν όλες ομαδοποιηθεί και θα βρίσκονται πια στο κτίριο CAD. Θα δείτε όμως απ' την άλλη ότι το σημαντικότερο τμήμα του προϋπολογισμού της αφορά τρέχουσες ταπάνες και σε πολύ μικρότερο βαθμό επενδύσεις, που είναι 6,7% του συνολικού προϋπολογισμού. Οι επενδύσεις αυτές ε, στόχο έχουν ώστε η ΓΑΜΑ το 2020 να έχει προβεί σε εξοικονόμηση και σε μείωση κατά 15% των δαπανών. Διότι το 2020 είναι η χρονιά όπου το σχέδιο αναδιοργάνωσης των υποδομών ασφαλείας και του εξοπλισμού ασφαλείας, όπως αποφάσισε το Προεδρείο του 2015, θα έχει ολοκληρωθεί. Λίγη η υποθεσμία και είναι η τελευταία χρονιά επενδύσεων για την ανακαίνιση της, ε, των υποδομών στον τομέα της ασφάλειας και του εξοπλισμού ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο ολοκληρώσαμε λίγο πολύ ουσιαστικά ολοκληρώσαμε ε, τον εξοπλισμό ασφαλείας σε όλες τις εισόδου των κτηρίων, στις τρεις ε, τόπους εργασίας και, στις, ε, και στα πάρκινγκ και θα ξεκινήσουμε, έχουμε ξεκινήσει να αναπτύσσουμε και τα νέα μπάντζα, τις νέες κάρτες αυτές που θα είναι πολύ πιο ασφαλείς από τις σημερινές για την είσοδο στα κτίρια με την ε, βοήθεια της νέας ε, τεχνολογίας, της πιο τελευταίας, πιο σύγχρονης τεχνολογίας και για να αναφερθούν αυτά τα νέα badge θα αξιοποιήσουμε την προεκλογική περίοδο για να τα, τα δώσουμε σε όλους τους ε, υπαλλήλου και σε ό,τι αφορά τους νέους βοηθούς και τους νέους βουλευτές βέβαια αυτό θα γίνει άμα τη αφήξη του τον Ιούνιο. για την εκπαίδευση να μιλήσω εν συντομία αφότου προσλήφθηκαν υπάλληλοι για το τομέα της ασφάλειας στο Κοινοβούλιο, άρχισε και η πολιτική εκπαίδευση ε, υψηλού επίπεδου. Για να είναι ο μεγαλύτερος δυνατό. Ε, να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερο δυνατό επαγγελματισμό των υπηρεσιών. Δέκα μέρε το χρόνο εκπαιδεύονται οι υπάλληλοι. Εν μέρη υποχρέωση ανακύκλωση. και εν μέρη εκπαίδευση ό,τι αφορά την εξέλιξη της ασφάλειας, όπως ε, παρατηρείται τον τελευταίο, τελευταίο καιρό. Σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, υπάρξε σήμερα Έχουμε, ε, είμαστε εντό χρονοδιαγράμματο Προεδρείου. Ξεκίνησε αυτό το project το 2015, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 2020. Και ο ενδεικτικό προπολογισμό τότε εκτιμούσε ήταν μεταξύ 25 και 30 εκατομμύρια τότε στο Προεδρείο. Νομίζω ότι εμείς θα ε, έχουμε τη ρίση την προθεσμία του 2020. Θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία του συναδέλφου που εργάστηκαν γι' αυτό και επίσης θα παραμείνουμε και στον προϋπολογισμό που θα είναι και πολύ κατώτερος μάλιστα αυτού που προβλεπόταν αρχικά. Κατά μέγιστο 22-23 εκατομμύρια θα δαπανίσουμε. Οι οικονομίες που κάναμε είναι γιατί κάναμε εσωτερικές μελέτες εδώ. Ε, επίσης, σε ό,τι αφορά ε, την προηγμένη τεχνολογία. Ε, είχαμε πολύ καλούς διαγωνισμούς ε, που έδωσαν καλό αποτέλεσμα για την υπηρεσιακή. Επίσης καταφέραμε να διατηρήσουμε εξοπλισμό συμβατό με τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσουμε. Όλα αυτά, όλες αυτές οι οικονομίες θα ήταν και πολύ μεγαλύτερες αν δεν χρειαζόταν να αντιμετωπίσουμε αύξηση της περιμέτρου κάτι που είδαμε τελευταία και ιδίως μετά τις επιθέσεις ε, στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες ε, και με τα έργα που έγιναν σε στενή συνεργασία με τη ΓΑΜΑ τα ΙΝΛΟ ε, χρειάστηκε να ενισχυθούν οι εισόδοι. τα σημεία ελέγχου είναι πολύ περισσότερα, όπως και τα σημεία πρόσβασης είναι πολύ περισσότερα. Παρά τη μεγάλη αυτή όμως αύξηση καταφέραμε να ελέγξουμε, να συγκρατήσουμε το κόστος. Αυτά είχα να πω για τον προπολογισμό. Και βεβαίω είμαι και στη διάθεσή σα να απαντήσω ευχαριστώ σε ερωτήσει σα. Ευχαριστώ. Many thanks, Mr. Uh, and also... Ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστώ γιατί μιλήσατε και λιγότερο από τον χρόνο μιλία που σα είχαμε κατάβα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στη Γενική Διεύθυνση Τραντ. Προηγουμένως η ε, ερωτήσει του εισηγητή και των σκιωδών. Έχω μία ερώτηση, λέει ο κύριος ε, Μάρκα, Μάνκα. Έχετε μεγάλη εμπειρία σαν ε, διευθυντής και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και από άλλα θεσμικά όργανα αυτή η τεχνογνωσία, αυτή η εμπειρία ίσως ε, μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε κάποιες εξοικονομήσεις. Βλέπετε σε αυτόν τον τομέα περιθώριο για περισσότερες εξοικονομήσεις και μείωση των δαπανών. Ο κύριος Ρούμπιχ, η δικό μου ερώτηση αφορά το θέμα της ε, προστασίας από την πυρκαγιά. Αναφερθήκατε σε αυτό. Θέλω να ξέρω αν οι ασκήσεις που γίνονται, εάν το θέμα των εξοπλισμών, εάν όλα αυτά που αναφέρατε προβλέπουν τον περιορισμό μιας ε, σημαντικής πυρκαγιάς. Θέλω να ξέρω αν ο εξοπλισμός που έχουμε είναι αξιόπιστος, γιατί μπορεί μια πυρκαγιά, όπως ξέρετε, να διαρκέσει μέχρι και δύο συνεχείς ημέρες, εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω φιλανδικά. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτήν την πάρα πολύ λεπτομερή παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί μας ενημερώσατε για την κτηριακή πολιτική. Εδώ στο κοινοβουλίο υπάρχει μια κατάσταση όπου δεν ενημερωνόμαστε πολύ για τα κτίρια. Είναι ένα πολύ σημαντικό όμω ποσό που διατίθεται σε αυτή την κτηριακή πολιτική. Θα ήθελα λοιπόν να έχω πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και τώρα μας τις παρουσιάσατε. Όσον αφορά το κτίριο ΣΠΑΚ, εδώ και χρόνια μιλάμε για το τι θα γίνει με το κτίριο αυτό και εκπλήσωμαι γιατί βλέπω ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για το τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί? Μα γιατί παίρνει τόσο χρόνο αυτή η απόφαση. Θα ήθελα να μου πείτε πιο συγκεκριμένα για τα 12 εκατομμύρια ευρώ Πού ακριβώς θα πάνε αυτά τα 12 εκατομμύρια, πού θα διατεθούν. Η δεύτερη ερώτησή μου, δεν ξέρω πώς να την εκφράσω, πώς να τη διατυπώσω. Η κακή συμπεριφορά, η κακή διαχείριση. Αυτά τα χρήματα κατανέμονται με σκοπό οι βοηθοί και οι ασκούμενοι, οι μαθητευόμενοι να εκπαιδεύονται. Μήπως ε, θα έπρεπε να στηρίξουμε όλους τους βοηθούς και τους ε, ασκούμενους με ένα καλύτερο τρόπο. Υπάρχουν, ε, αν θέλετε, και ψυχολόγοι, ψυχολογική υποστήριξη για περιπτώσεις παρενοχλήσεων. Θα πρέπει να έχουμε ειδικού, θα πρέπει να έχουμε κάποιους εμπειρογνώμονες για να μπορούν να επέμβουν όταν συμβαίνουν τέτοιες περιπτώσεις. Η κυρία Γιάτα Μάκε κάνει την ερώτηση αυτή, αλλά κυρία Γιάτα Μάκε, εδώ το θέμα μας είναι η ασφάλεια και στις 5 θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει χρόνος για τις τελευταίες ερωτήσεις. Δεν ξέρω σε ποια γενική διεύθυνση απευθυνόταν η τελευταία αυτή ερώτηση. Πάντως όχι στη ΣΕΙΦ και όχι στην Ίνλο. Ας απαντήσουμε όμως τις δύο πρώτες ερωτήσεις του κυρίου Μάνκα και του κυρίου Ρουμπίκ και θα δούμε αν έχουμε χρόνο για τελευταία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι όσον αφορά την ασφάλεια πολλές φορές φαίνεται δύσκολο να υπάρξει συνέργεια μεταξύ των θεσμικών οργάνων, μεταξύ των ε, θεσμών, καθότι ο κάθε ένας είναι πολύ εξειδικευμένος, με πολλές ιδιαιτερότητες. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ στο Κοινοβούλιο δεν είναι οι ίδιες ε, απαιτήσεις ασφάλειας που προκύπτουν στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, ίσως και επειδή έχει αλλάξει η κατάσταση και υπήρξαν αυτά τα πρόσφατα γεγονότα, συνεργαζόμαστε πολύ περισσότερο μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Κύριε Μάνκα, και όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες για όλες τις αποστολές που κάνουν οι αντιπροσωπείς μας στο κόσμο. Δεν δαπανώνται υπέρογκα ποσά για να εντοπιστούν τα στοιχεία και οι πληροφορίες που χρειαζόμαστε, αλλά απευθυνόμαστε εκεί που υπάρχουν, εάν υπάρχουν σε ένα άλλο θεσμικό όργανο. Έχουμε συμβόλαια και συμβάσεις με την Επιτροπή 30 διαφορετικά γραφεία με τους οποίους συνεργαζόμαστε με την ε, Επιτροπή. Έχουμε μία υπηρεσία φύλαξης και έχουμε εξοικονομήσει πολύ σημαντικά ποσά και εμείς και η Επιτροπή και πολύ λιγότερη γραφειοκρατία. Συνεργαζόμαστε επίσης στενά και με όλα τα άλλα θεσμικά όργανα, με μεγάλη επιτυχία θα έλεγα, παραδείγματος χάρη από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και πέρα οι συνάδελφοι υπάλληλοι μπορούν να έρθουν εδώ στο Κοινοβούλιο χωρίς να περάσουν από έλεγχο ασφάλειας. Μπορούν να πάνε στην Επιτροπή των Περιφερειών, στο δικαστήριο με άμεση αναγνώριση του μπάτζ. Δεν χρειάζεται δηλαδή ειδικό έλεγχος. Σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο badge και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα πρέπει να εναρμονιστεί η διαδικασία για την ε, διαπίστευση, αυτή δηλαδή που ισχύει στα τρία θεσμικά όργανα. Τα κτίρια μας είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Οι συνάδελφοι του Κοινοβουλίου μπορούν να πάνε με εσωτερική διάβαση στην Επιτροπή των Περιφερειών χωρίς να βγουν έξω. Συνεργαζόμαστε λοιπόν στενά σε θέματα ασφάλειας. Πολλές φορές βεβαίως, επαναλαμβάνω κάτι που ήδη είπα, εξαιτίας των ε, συμβάντων στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας έχει αλλάξει ριζικά. Η ασφάλεια λοιπόν έχει αλλάξει, τα μέτρα ασφάλειας έχουν αλλάξει και ο καθένας από εμά απευθυνόταν στο παρελθόν στις αρχές του Βελγίου, του Λουξεμβούργου και της Γαλλίας και ο καθένας προσπαθούσε να λύσει μόνος του τα προβλήματα ασφάλειας που αντιμετώπιζε. Από το 2014 οι τρεις πρόεδροι των θεσμικών οργάτων συνεργάζονται και απευθυνόμαστε με έναν ενιαίο τρόπο στις αρχές των κρατών μελών. Αυτό μας διευκολύνει, υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των ε, υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας. Το θέμα των χώρων στάθμευσης, η πρόσβαση στα κτίρια και τα θέματα προστασίας, πυρασφάλειας και η συγκεκριμένη προστασία και εξοπλισμοί που υπάρχουν στα κτίρια μας είναι αντικείμενο επανοργάνωσης. Οι χώροι στάθμευσης ε, είναι σε φάση πλήρους ε, αναδιοργάνωσης με σκοπό να αυξηθεί η ασφάλεια. Μια κοινή ομάδα εργασίας για την ασφάλεια και τα κτίρια έχει ολοκληρώσει την ε, εργασία της και αρχές Μαρτίου θα είμαστε σε θέση να υποβάλουμε τα πρώτα πορίσματα και το Προεδρείο θα μπορεί να αποφασίσει πριν το τέλος της θυσίας. Κυρία Γιατάκη, δεν κατάλαβα γιατί απευθύνατε σε μένα την ερώτησή σας. Μάλλον στην κυρία Λίνους πρέπει να την απευθύνετε. Είναι μάλλον αρμόδια και ίσως να μπορεί και να σας απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Καρότσα. Έχουμε λίγα λεπτά με την Γενική Διεύθυνση SAFE. Πότε μπορούμε να περιμένουμε αμοιβαιότητα όσον αφορά τους ελέγχους των μελών του Κοινοβουλίου που επιθυμούν να μπουν στα κτίρια του Συμβουλίου. Πολύ περίπλοκο το θέμα αυτό. Εμείς ήμασταν ε, οι πρώτοι που προτείναμε με το Δικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν έχουμε ακόμα πετύχει αυτή την συνεργασία με το Συμβούλιο. Ξέρετε ότι το Συμβούλιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια. Έχουν πραγματικά δημιουργήσει ένα φρούριο, ένα μπούνκερ και προς το παρόν δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι τέτοιο. Αλλά συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ίσως όχι με γενικευμένο τρόπο όπως το κάναμε με την Επιτροπή και τους άλλους θεσμούς, αλλά ενδεχομένως εν μέρη πρόσβαση θα μπορούν να έχουν τα μέλη του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο. Ναι, εγώ πραγματικά εκπλήσωμαι που το Συμβούλιο έχει θωρακιστεί και έχει θωρακίσει τα κτίρια του σαν φρούρια τόσο πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα και ενδεχομένω θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό αν μας μείνει χρόνος. Η Γενική Διεύθυνση Τραντ, ο κύριος Βάλτερ Μαύριτς, έχει το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να συνομιλήσω με εσά, τον εισηγητή την κύριο Μάνκα και του συγκεκριμένου συναδέλφου. Μοναδική ευκαιρία να μιλήσουμε για τις μεταφραστικέ υπηρεσίες και τι μας οδήγησε να ζητήσουμε αυτό που ζητήσαμε για τον προπολογισμό του 2020. Ο κ. Κεντή ε, εξήγησε πολύ καλά τις ε, αρχές και τις κατευθυντήρες γραμμές που ακολουθήθηκαν για τα διάφορα αιτήματα που υποβάλαμε. Συμμορφωθήκαμε με τις αρχές. Θελήσαμε να δούμε ποια είναι η αποστολή της Γενικής ε, του, του μεταφραστικού μετάφρασης, ποια είναι η αποστολή και ποια είναι, τα, ποια είναι η πρικοδότηση που έχουμε και τα μέσα που διαθέτουμε. Η αποστολή φαίνεται απλή θεωρητικά, αλλά στην υλοποίηση είναι περίπλοκη. Ποια είναι η αποστολή να μεταφράζουμε, να προσαρμόζουμε και να μεταφράζουμε ή να μεταδημιουργούμε σχεδόν τα πάντα τα οποία έχουν γραφτεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκτός Ευρωκοινοβουλίου, κυρίως όταν μιλάμε για συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ετοιμάζουμε πολυγλωσσικά προϊόντα, τα οποία διαβιβάζονται πηγαίνουν κυρίως στους ευρωβουλευτές αλλά απευθύνονται και στους πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προϊόντα μας άμεσα ή έμεσα. Αυτές είναι οι αποστολές της μεταφραστικής υπηρεσίας και γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποια στήριξη. Ε, χρειαζόμαστε προσωπικό, Φερρυπίν. Βασικό στοιχείο. Είμαστε η μεγαλύτερη υπηρεσία, η μεγαλύτερη γενική διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε περίπου 1.200 ε, που είναι το προσωπικό μας. Οι περισσότεροι βρίσκονται στο Λουξεμβούργο. Οι περισσότεροι είναι μεταφραστές και μεταφράστριες. Αλλά όχι μόνο αυτό. Έχουμε και άλλες ειδικότητες που εργάζονται στη μετάφραση. Αυτή η ανάγκη μας λαμβάνεται υπόψη και στην κατάρτιση του προπολογισμού. Θα αναφερθώ αργότερα σε αυτό. Να ευχαριστήσω σε αυτό το στάδιο πολύ θερμά το προσωπικό της Γενικής Διευθύνσεως Μετάφρασης, κυρίως τώρα προς το τέλος της θητείας. λάβαμε υπόψη τις αρχές που καθορίστηκαν, όπως σας είπα. Λάβαμε υπόψη τους στόχους μας και τα μέσα που έχουμε στη διαθέσή μας. Σε τρεις τομείς έχουμε ανάγκες. Θέλουμε πρώτα απ' όλα να έχουμε αποδοτικότητα στον αφορά χρήση των πόρων. Μετά θέλουμε να είμαστε καινοτόμοι. Και τρίτον θέλουμε να συμμορφωνόμαστε με καλές προδιαγραφές για την αποδοτική χρήση των πόρων. Πρώτος στόχος. Όλοι ξέρουν ότι βλέπουμε πόσο παράγουμε, πόσο εργαζόμεθα και πόσο αποτελεσματικοί είμαστε στην εργασία μας. Αυτή η γραμμή αναφέρεται και στη βοήθεια που παίρνουμε απ' έξω, από τους εταίρους μας, που μας βοηθούν Το 2018, παραδείγματο χάρη, είχαμε παράγει 2,7 εκατομμύρια σελίδες. Η εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών αναλογεί στο 30% της ε, εργασίας μας. Και αυτή η εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών θα μας κόστιζε 8,2 εκατομμύρια ευρώ. έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα ε, δημόσιας ανάθεσης, διαγωνισμών. Ε, και εκεί προσπαθούμε να καλύψουμε τις ποιοτικέ μας ανάγκες όσον αφορά τις μεταφράσεις. Αυτή είναι η βασική μας μέρημνα. Διότι θεωρούμε ότι είμαστε η καλύτερη μεταφραστική υπηρεσία στον κόσμο και γι' αυτό έχουμε μεγάλες απαιτήσει. Δημιουργήσαμε ένα νέο σύστημα που δρομολογείται πιστοποίησης εκείνων που θα συνεργαστούν μαζί μας, εξωτερικούς συνεργάτες. Η αποδοτικότητά μας εξετάζεται και σε συνάρτηση με την καινοτομία. Θέλουμε τεχνολογική καινοτομία που χρησιμοποιείται εντός της υπηρεσίας αλλά και διοργανικά και παίρνουμε τα μηχανήματα που είναι εμπορικά διαθέσιμα. Γλωσσική τεχνολογία ό,τι μπορεί να υποστηρίξει τη μετάφραση χρησιμοποιείται. Θέλουμε να είμαστε όμως και αποδοτικοί, να δίνουμε νέες υπηρεσίες που ζητεί το Κοινοβούλιο, που ζητούν τα μέλη και οι πολίτες. Σαφή διατύπωση, καθαρή γλώσσα. Μια γλώσσα εύληπτη για τους πολίτες να χρησιμοποιούμε. Τρίτος τομέας. Δεύτερος τομέα, συγγνώμη. Είναι 6,2 εκατομμύρια ευρώ. Κοστίζει. Αυτά είναι τα δύο βασικά κονδύλια του προπολογισμού. Ο τρίτο τομέα που χρηματοδοτείται αποτελείται από δύο γραμμέ του προπολογισμού σχετίζονται με τα επαγγελματικά πρότυπα, τι επαγγελματικέ προδιαγραφέ που θέλουμε να χρησιμοποιούμε στην μετάφραση, στην πολυγλωσία. Είμαστε μία από τι καλύτερε μεταφραστικέ υπηρεσίε στον κόσμο. Πολλοί μα έχουν σαν παράδειγμα. Θεωρούμε ότι ηγούμεθα σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα. Υπέχουμε καθήκον να συμμετέχουμε και στον καθορισμό των προτύπων, έτσι το βλέπουμε. Χρειαζόμαστε συνεργασία με πανεπιστήμια, συστήματα μαθητείας, εκπαίδευση του προσωπικού μας και να μοιραζόμαστε με τον υπόλοιπο κόσμο τις γνώσεις μας. 293.000 ευρώ χρησιμοποιούμε αυτό το σκοπό. Έχουν προγραμματίσει. Τέσσερα λοιπόν τα βασικά σημεία, οι βασικοί τομείς, συνολικά 14,9 εκατομμύρια ευρώ. Για την παροχή έξοχων υπηρεσιών, άκρο ποιοτικών και στηρίζοντα και την πολυγλωσία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Μαύρη. Ο εισηγητής όχι, ο κύριος Ρούμπικ όχι, κύριε Καρθιαθάμπαλ όχι. Να ρωτήσω εγώ τότε κύριε Μαύριτς. γιατί ήδη στα τέλη του 2018 εγκρίναμε μια μεταφορά πίστοσης για την ενίσχυση της υπηρεσία κατά 3 εκατομμύρια, συγκεκριμένα τους συμβασιούχους. Ο λόγος ήταν το αυξημένος φόρτος εργασίας που περιμένετε μέχρι τις εκλογές. Τώρα, στο σχέδιο των εκτιμήσεων για το 2020 αναφέρεται πάλι σημαντική αύξηση για τη γάμα δελτα τραντ. 58% αύξηση σε σχέση με το 19 για τους συμβασιούχους. Διαρωτώ με. Αν μπορείτε να μας δώσετε μια περαιτέρω εξήγηση για την ανάγκη αυτής της αύξησης. Γιατί φαντάζεται κανείς ότι στην αρχή της νέας θητείας ο φόρτος εργασίας στην δική σας γενική δεύση θα είναι λιγότερος, μικρότερος από ότι στο τέλος μιας Είναι λογικό αυτό που λέω αν θέλετε να μας εξηγήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την ερώτηση αυτή. Αυτό που θα θέλαμε είναι ο προπολογισμό για την εξωτερική ανάθεση μεταφράσεων μέσω είτε γραφείων μεταφραστικών είτε ιδιωτών να έχει κυκλικό χαρακτήρα. Όλο το σχεδιασμό μας από το έτος των εκλογών μέχρι τις επόμενες εκλογές. Έτσι τον αντιλαμβανόμαστε. Και πέρσι είχαμε τη μεγαλύτερη εχμή. Το πικ της νομοθετικής περίοδου. Λόγω και του ε, πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, των εγγράφων, ε, της νομοθεσίας της σχετικής. Επομένως, γι' αυτό χρειάστηκε να ζητήσουμε αύξηση του πολιτισμού που είχε μειωθεί στην αρχή του έτους. Αυτό το 18. Το 19 έχουμε 5 εκατομμύρια προπολογισμό ο σχέδιο, διότι κατά κύριο λόγο θα ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του νομοθετικού έργου τον Απρίλιο και δεν αναμένουμε μεγάλη αύξηση μέχρι όταν αναλάβει καθήκοντα νέα κομισιόν, άρα μιλάμε για Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2019. Γι' αυτό το 19 ζητάμε 5 εκατομμύρια. Όμως το επόμενο έτος, το 2020, προβλέπουμε κανονικό νομοθετικό έργο. Άρα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ το υπολογίζουμε. Και το ίδιο θα ισχύει και για το 2021 και για το 2022. Οπότε και περνάμε ξανά προς το τέλος της προσεχούς πλέον ε, κοινοβουλευτικής θητείας, όπου θα έχουμε πάλι αύξηση στο ε, τελευταίο έτος και το 2023-2024 θα έχουμε ένα διαφορετικό κύκλο νομοθετικού έργου. Και αυτό θα αντικατοπτρίζει και την εξωτερική ανάθεση. Θέλουμε πρώτα να καλύψουμε με εσωτερικού πόρου και μετά να προβούμε σε εξωτερικέ αναθέσει. Αυτή είναι η λογική μα. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ, κύριε. Γίνει και ο κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ. Ακούστε, κάθε θεσμικό όργανο και η μεταφραστική υπηρεσία, η υπηρεσία δερμηνίας έχει περίοδο εχμής, πίξ, Όπω είπε και ο γενικό διευθυντή, Τώρα, είναι τώρα πώς συμπεριφερόμαστε σε ε, μια τέτοια περίοδο εχμής. Ε, στρεφόμαστε σε κάποιο εξωτερικό συνεργάτη ή κοιτάμε δεξιά και αριστερά για να δούμε μήπως κάποιο άλλο θεσμικό όργανο θα είχε ε, στη διάθεσή του κάποια άτομα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Αφού έχουμε ένα πακέτο, αν θέλετε, είμαστε ένα πακέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα μήπως μπορούμε έτσι να προβούμε σε κάποιες οικονομίες και το δεύτερο είναι συνέργειες και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Thank you very much, Mr. Manka. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάνκα. Θα απαντήσω και στα δυο σας ερωτήματα με μία απάντηση. Η διοργανική συνεργασία είναι εντατική μεταξύ των μεταφραστικών υπηρεσιών. Και την έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό. Εγώ ήρθα το 2004 στο Κοινοβούλιο και ήδη τότε υπήρχε συνεργασία. Η συνεργασία έχει να κάνει κυρίως με τον τομέα της πληροφορικής, γιατί πιστεύουμε ότι η αποδοτική χρήση των πόρων μπορεί να γίνει και με την πολύ καλή χρήση της τεχνολογίας. Έχουμε λοιπόν αναπτύξει πολύ ξεκάθαρα κοινά πρότυπα στην πληροφορική ένα είδος ε, νέφους που μπορεί να μην είναι ακριβώ έτσι. Τέλο πάντων, είναι ένα iCloud στο οποίο αποθηκεύονται οι μεταφράσει. Όλε οι μνήμε αποθηκεύονται εκεί, σε αυτό το νέφο. Οπότε, όποτε χρειάζεται μια μετάφραση από παλιότερα, πηγαίνουμε σε αυτό το νέφο να την αναζητήσουμε, που είναι κοινό το νέφο για όλα τα θεσμικά όργανα. Ε, πληρώνουμε περίπου 700.000 ευρώ για την ε, δημιουργία ολοκλήρωση αυτών των κύκλων ε, και συνεργαζόμαστε πολύ καλά ώστε όλοι να εξοικονομούμε πόρους και να καινοτομούμε ταυτόχρονα. Δεν σταματάμε όμως εκεί. Έχουμε επίσης αναπτύξει και ένα σύστημα, μια πλατφόρμα που λέγεται Workload Balancing System. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε και εσείς. Όποτε κύριε Μάνκα υπάρχει ε, κάποια ε, δυνατότητα να αξιοποιήσουν προσωπικό από άλλα θεσμικά να Το είδαμε αυτό και στο πολιτές σαμικό πλαίσιο. Ακόμα και πριν κάνουμε ένα εξωτερική ανάθεση, στρεφόμαστε στην πλατφόρμα αρχικά και ε, ζητούμε μήπως υπάρχουν διαθέσιμοι από άλλα θεσμικά όργανα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Βέβαια όλοι ήμασταν πάρα πολύ απασχολημένοι και ταυτόχρονα, οπότε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν δύσκολα. Αλλά υπάρχει αυτή η πλατφόρμα ε, που είναι στο επίπεδο των γλωσσικών κοινοτήτων ε, και κάθε ε, γλωσσική κοινότητα συνεργάζεται. Η συνέργεια, συνεργασία πηγαίνει στον τομέα των ανθρώπινων πόρων επίσης, ιδίως όταν συνδυάζουμε και σχεδιάζουμε για το μέλλον, τα προφίλ που θα χρειαστούμε, πώς θα εξελιχθεί το επάγγελμα, τι είδους υπηρεσίες θα έχουμε να παράσχουμε στον τομέα της πολυγλωσσίας και με τους διαγωνισμούς μας ε, στο πλαίσιο έψο. Επίσης ε, προσλαμβάνουμε και κόσμο. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Um, that ends, uh, Ευχαριστώ κύριε Μαύριτς. Τελείωσε λοιπόν η συζήτηση με την Γενική Διεύθυνση ΤΡΑΤ και τέλος εξίσου σημαντική η Γενική Διεύθυνση ΛΙΝΚ. Η κυρία Αγνέσκα Βάλτερ Ντρόπ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι είμαστε μια ομάδα εδώ. Χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να ανταλλάξω μαζί σας κάποιες απόψεις κλείνοντας την ακρόαση. Μοναδική ευκαιρία για μένα και για τους συναδέλφους να παρουσιάσω τις, τα αιτήματά μας για τον προπολογισμό του 2020 και να παρουσιάσω το πλαίσιο των εργασιών που κάνουμε και των υπηρεσιών που παρέχουμε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του Ευρωβουλευτές. Η Γενική Διεύθυνση Link, η Γενική Διεύθυνση για Επιμελητία και Διερμηνία για Διασκέψεις είναι υπεύθυνη για γλωσσική υποστήριξη, τεχνική διοργάνωση, γενική υποστήριξη των συνεδριάσεων και διασκέψεων. Αναδιορθωθήκαμε πρόσφατα. Έχουμε νέο όνομα και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα απόφασης του Προεδρείου του Δεκεμβρίου του 2017 όσον αφορά τη στρατηγική εξυγχωρισμού της διαχειρίσεως των διασκέψεων και συνεδριάσεων έδωσε στο Γενικό Γραμματέα το Προεδρείο και εκείνος μας έδωσε εντολή να αναπτύξουμε μια σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά την εξυπηρέτηση των συνεδριάσεων και των εκδηλώσεων στο Κοινοβούλιο βασιστήκαμε στην ε, καλή παράδοση που υπήρχε και τις υπηρεσίες ε, που ήδη ε, χρησιμοποιούσαμε. Συμπεριλάβαμε και το θέμα της οργάνωσης των συνεδριάσεων, της υποστήριξης των συνεδριάσεων. Έχουμε και τους κλητήρες μαζί μας, τους τεχνικούς των διασκέψεων, την τεχνική υποστήριξη που παρέχεται στις συνεδριάσεις. Αλλά βέβαια έχουμε και πασίγνωστη υπηρεσία των ε, διερμηνέων συνεδριάσεων που παρέχουν έξοχες υπηρεσίες και που είναι παρόντες σε αυτή τη συνεδρίαση. Δεν θα επισέθω λεπτομέρειες όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Ε, είμαστε περίπου στα, ε, στα μισά όσον αφορά το μέγεθος Γενικής Διευθύνσεως και εκπληρώνουμε την αποστολή της υποστηρίξεως της πολυγλωσσίας. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο κονδύλι υποστήριξης πολυγλωσσίας. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ εκτενέστερα στην πτυχή των συνεδρίων, της διοργάνωση των συνεδρίων, διότι πιστεύω ότι αυτό ήταν κάτι σχετικά, ήταν κάτι καινούριο, πολύ ενδιαφέρον Εγχείρημα που απαιτεί όμως και περισσότερη οικονομική υποστήριξη. Άρα και ανάγκες για τον προπολογισμό. Τούτου λεχθέντος, αυτό που είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη είναι ότι θέλουμε να επετύχουμε οικονομία κλίμακας να έχουμε καλύτερη διαχείριση τη στήριξη των διαφόρων παρεχομένων υπηρεσιών. Υπηρεσιών που στηρίζουν τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και διαφόρων εκδηλώσεων του Κοινοβουλίου. Ε, που αυτέ οι εκδηλώσει είναι διάσπαρτε στο Κοινοβούλιο και συνεδριάσει. Θέλουμε να έχουμε ένα σημείο επαφή για εκείνου που θέλουν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίε ε, συνεδρίων, να παρέχουμε ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη και να βοηθήσουμε αυτούς που θέλουν να διοργανώσουν τις συναντήσεις και διάφορες και συναντήσεις όπως είναι η συνεδριά των επιτροπών. Ξεκινήσαμε να το πραγματοποιούμε αυτό. Αυτή την υπηρεσία την παρέχουμε εδώ και χρόνια για τις πολιτικές ομάδες, για συνεδριάσεις εκτών των τριών εδρών του Κοινοβουλίου και έχουμε αναπτύξει τέτοια ολιστική υπηρεσία και για διασκέψη ψηλού επίπεδου κάτι που διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του 2018 και του 2019 για διακοινοβουλευτικέ συνεδριάσεις, για συνεδριάσεις αντιπροσωπιών. Τώρα θέλουμε να δούμε πώς θα διευρύνουμε το πλαίσιο, να καλύπτουμε και εκδηλώσεις ε, στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά υπάρχουν και δυνατότητες να προχωρήσουμε πιο πέρα όσον αφορά τη συνεργασία και να απευθυνθούμε, να ανοιχτούμε προς την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και θα προσπαθήσω να καλύψω και κάποια σημεία που ανέφερε ο κύριος Μάνκα σε λίγο. Θέλουμε να βρούμε νέα εργαλεία, καινοτόμα εργαλεία, που θα χρησιμοποιήσουμε. Ξεκινήσαμε ήδη ένα πρόγραμμα για να δώσουμε στο Κοινοβούλιο ένα εργαλείο καταχώρησης των συμμετεχόντων, το Regis. Και είμαι σίγουρη ότι όλοι θα μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτό, όχι μόνο οι οργανωτές διαφόρων συνεδριάσεων, αλλά θα ωφεληθούν και οι ευρωβουλευτές, αλλά και διάφορες υπηρεσίες. Και είμαστε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση SAFE, για να βελτιώσουμε και τις συνθήκες ασφαλείας εντός του Κοινοβουλίου μέσω του Μητρώου αυτού, των συμμετεχόντων. Θέλουμε να το επεκτείνουμε αυτό το σύστημα στο μέλλον. διότι έχουμε ανοιχτεί και προς τις δύο, έχουμε διασυνέσεις με τις δύο επιτροπές, μπορούμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις αυτές περαιτέρω θέλουμε να βρούμε και άλλα καινοτόμα μέσα υποστηρίξεως των συνεδρίων. Ελπίζω το νέο κοινοβούλιο να έχει κάποια προσφορά, νέα προσφορά, να έχουμε μια εφαρμογή για τους συμμετέχοντες, εφαρμογή για το τηλέφωνο, ένα app, θα μπορεί να τους διευκολύνει να βρίσκουν έγγραφα και θα τους παρέχει και κάποια βοήθεια και υποστήριξη κατά διάρκεια των συνεδριάσεων. είναι εξοικονομήσει σε δύο επίπεδα πετυχαίνουμε. Δηλαδή, συναθρίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και απελευθερώνουμε πόρους για άλλες γενικές διευθύνσεις, αναλαμβάνοντας κάποια καθήκοντα. Η DG-Link είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των εκθέσεων των μελών, τη σχετική υπηρεσία, και αναλάβαμε και τη διοργάνωση των, οργανώσ... εκδηλώσεων στην πλατεία, στην Εσπλανάτ. Ό,τι σχετίζεται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων στι αίθουσες συνεδριάσεων στο εσωτερικό χώρο, η σχετική υποστήριξη καλύπτεται από εμά. Θέλουμε να δούμε πώ θα διαχειριστούμε καλύτερα όλα αυτά και πώ οι διαδικασίε θα εξομαλυνθούν, θα γίνουν πιο ευέλικτε και θα έχουμε και υποστήριξη μέσω ενία στηρίδας. Θα χρησιμοποιούμε και τη σχετική τεχνολογία. Εδώ και χρόνια ανανεώνουμε τις αίθουσες συνεδριάσεων, συνεχής αένα η διαδικασία, ανακαίνιση αυτών. Έχουμε 100 αίθουσες συνεδριάσεων περίπου στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Συμπεριλαμβανομένων και των καμπινών διερμηνίας, ό,τι σχετίζεται με τον ήχο, όλα αυτά τα καλύπτουμε εμείς Συνεργαζόμαστε με τη Γενική Διεύθυνση Ίνλο και τη Γενική Διεύθυνση ΚΟΜ και με την ITEC για να έχουμε σφαιρική ολιστική προσέγγιση και να έχουμε οθόνες που να χρησιμοποιούνται πολλαπλώς και για βιντεοδιασκέψεις και για παρουσιάσεις, να έχουν πολλαπλές χρήσεις οι οθόνες, οι οθόνες κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Αναπτύσσουμε επίσης εργαλεία με προθυμένη τεχνολογία, προχωρημένης τεχνολογίας για ψηφιακή σήμανση στο Κοινοβούλιο και καθοδήγηση ηλεκτρονικά, ε, ηλεκτρονικές αφήσει ή πόστερ. Προσπαθούμε να τα ψηφιοποιήσουμε όλα για την ε, στήριξη των εκδηλώσεων και των διασκέψεων και των συνεδρίων. Όλα αυτά απαιτούν πρόσθετες επενδύσεις. Γι' αυτό ζητάμε χρήματα σε, τρία, σε τρεις γραμμές του προπολογισμού. Έχουμε αύξηση, ζητάμε αύξηση περίπου κατά 11 εκατομμύρια ευρώ που θα διατεθούν για αυτούς τους σκοπούς που ανέφερα. Άλλο θέμα που έχω ήδη αναφέρει και το αναφέρω εκ νέου είναι η διερμηνία συνεδρίων. Όπως είπα, Βασιζόμαστε στις έξοχες υπηρεσίες που παρέχει, παρέχουν, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε με τον καιρό και να προσαρμοστούμε τις ανάγκες του θεσμικού οργάνου. Στον τομέα της Ερμήνειας, βασικός στόχος ήταν αυτός της διαδικασία αλλαγής των συνθήκων εργασίας των διερμηνέων. Μετά από 4,5 χρόνια ολοκληρώθηκε όλη η διεργασία αλλαγής συνθήκων εργασίων πέρσι και μπορέσαμε να έχουμε ένα πλαίσιο τώρα, το οποίο πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρουμε περισσότερο χρόνο συνεδριάσεων σε πολυγλωσσικές συνεδριάσεις στο Κοινοβούλιο. Πρώτα παραδείγματα που μου έρχονται στο νου. Έχουμε προσφέρει στο Κοινοβούλιο, κυρίως στις Επιτροπές αλλά και σε άλλους φορείς, περισσότερο χρόνο συνεδριάσεων, επιτρέποντας συνεδριάσεις τεσσάρων ωρών χωρίς συμπληρωματικό κόστος, χάρη στις νέες συνθήκες εργασίας των διερμηνέων και ότι ε, πάνω από 50% των ε, συνεδριάσεων στο Κοινοβούλιο είναι βραχύτερε από δύο ώρε και μπορούμε να διαθέτουμε διερμηνεί. Πριν από 15 χρόνια, περισσότερε συνεδριάσει διαρκούσαν 3,5 ώρε. Και όλε αυτέ οι συνεδριάσει διάσπαρτε κατά τη διάρκεια τη ημέρα σε διάφορε χρονοθυρίδε και μπορούμε αυτό να το κάνουμε, να έχουμε την κάλυψη με νέε συνθήκε εργασία χωρί να έχουμε πρόσθετε προσλήψει. Έχουμε αυτή τη συμφωνία για τις συνθήκες εργασίας που υποστήριξαν όλα τα μέρη και οι εκπρόσωποι των διερμηνέων και λάβαμε υπόψη τα θεμητά ε, δικαιώματα των διερμηνέων και τις ανάγκες συμφιλίωσης ιδιωτικής ζωής με εργασία. Όλα αυτά ελήφθησαν υπόψη στο νέο πλαίσιο. Τούτου λεχθέντος βλέπουμε μπορούμε να καλύπτουμε περισσότερες συνεδριάσεις το 2018 Είδαμε τριπλάσιες ε, συνεδριάσεις τεσσάρων ώρων από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Οι επιτροπές λοιπόν και διάφοροι φορείς χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει μια ανάγκη για περισσότερο χρόνο συνεδριάσεων και βλέπουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες ε, αλλά αξιολογήσαμε και τις ανάγκες για την 1405 του προπολογισμού για εξωτερική ανάθεση διερμηνίας παρέχουμε διερμηνία σε μεικτό μοντέλο. Έχουμε συναδέλφους που έχουμε εδώ, σήμερα εδώ παρόντες, ανήκουν, είναι και μέλη του προσωπικού που είναι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου, καθώς και ελεύθερες επαγγελματίες που είναι συμβασιούχοι, είναι freelance. Έτσι, δημιουργεί, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Εργάζονται από κοινού οι συνάδελφοι σε μια ομάδα και παρέχουν ε, ποιότητα, ποιοτικές υπηρεσίες. αξιολογούμε τις συνέπειες των νέων συνθήκων εργασία. Χρειάζεται χρόνο να εξετάσουμε τον πλήρη αντίκτυπο των νέων συνθήκων. Το πρώτο αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι ότι παρέχουν περισσότερε υπηρεσίε, μπορούν να παρέχουν περισσότερε υπηρεσίε, αλλά θεωρούμε ότι ίσω χρειαστούμε και λιγότερου πόρου. Μία μείωση 3,6% σε αυτή τη γραμμή σε σχέση με το 2018, που είναι η περίοδο σύγκριση για μα. Το 2019 το, η δραστηριότητά μας αναμένεται να μειωθεί. Ε, κάθε εκλογικό έτος ζητούμε ένα ποσό και τελικά καταναλώνουμε λιγότερα χρήματα από το ποσό που ζητήσαμε από αυτό το κονδύλι. Συνεργαζόμαστε επίσης με τις άλλες υπηρεσίες διερμηνίας άλλων θεσμικών οργάνων για να πετύχουμε οικονομία κλίμακας. Κυρίως το τέλος όσον αφορά τις προσλήψεις και πληρωμές των freelance και τη διαπίστευση αυτών. Αυτό γινόταν και γίνεται ήδη. Αλλά απαντώντας στον κύριο Μάνκε, να, ήθελα να πω ότι παρέχουν υπηρεσίε και σε άλλα θεσμικά όργανα και τις συμβουλευτικέ επιτροπές. Κατά αποκλειστικότητα εργαζόμαστε για το συνήγορο του πολίτη, για το ελεκτικό συνέδριο και βλέπουμε τώρα με τις νέες συνθήκες εργασίας κυρίως με τη, η, ΟΚΕ, η ΕΟΚΕ, έχει αυξήσει τις παραγγελίες της εντός εισαγωγικών και βλέπουμε ε, περιθώριο για αύξηση της συνεργασίας και περισσότερες οικονομίες κλίμακας. Επίσης θα έλεγα ότι σίγουρα γενικότερα με την ευρύτερα έννοια της υποστήριξης συνεδρίων θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία. Οι αίθουσε συνεδριάσεων είναι κοντά η μία στην άλλη. Ήδη διαθέτουμε στι επιτροπέ τα εργαλεία πληροφορική για κρατήσει. Διευκολύνονται έτσι και μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα. Αν δείτε τις επενδύσεις, όταν κάνουμε τις ανακαινήσεις των αιθουσών, θα δούμε μήπως μα συμπεριλάβουμε να καλύψουμε τις ανάγκες για τεχνική διαχείριση, ε, αλλαγή του εξοπλισμού. Αυτό ίσως να είναι εποφελές ε, για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τώρα είναι διαφορετικά κονδύλια. Πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπών που ισχύει από το 2014, αν δεν κάνω λάθος. Εν κατακλείδη, αυτά έχω να πω. Ζητώ συγγνώμη που χρονοτρίβησα, αλλά είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Walter Ο κύριος Μάνκα, ο εισηγητής. Αρχικά είχατε μία ερώτηση για την DigiLink όσον αφορά το κόστος Θέλετε κάποιες διευκρινήσεις για την επεξήγηση ψήφου και το κόστος αυτής της διαδικασίας. Έχετε και άλλες ερωτήσεις. Ναι, έκανα αυτή την ερώτηση. Είναι όμως πολιτικό το θέμα, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η αξιολόγηση, ποιο είναι το κόστος. Μπορεί να μην την έχετε την απάντηση σήμερα. Αλλά πόσο ακριβώς στοιχίζει αυτή η διαδικασία επεξήγησης ψήφου. Οι σκιώδεις αποφάσισαν ότι οι επεξηγήσεις ψήφου θα πρέπει να μην γίνονται με αυτόν τον τρόπο, να αλλάξουμε τη διαδικασία, δεν είναι αποτελεσματική. Προσπαθούμε λοιπόν να ξαναδούμε αυτή τη διαδικασία, αλλά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ποιο είναι το κόστος της διερμηνίας. Πόσο στοιχίζει η επεξήγηση ψήφου. Ίσως και στη Γενική Διεύθυνση Finance μπορούμε να κάνουμε την ίδια ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ να σας δώσω την απάντηση αμέσως αλλά κάναμε μια γενικότερη, αν θέλετε, αξιολόγηση, χοντρικά. Προσπαθήσαμε δηλαδή να δούμε τι ανήκει στην επεξήγηση ψήφου και τι μπορεί να μπει σε άλλες κατηγορίες ε, σε μια συνεδρίαση της Ολομέλειας. Έχουμε λοιπόν κάποια τιμή, αν θέλετε, που μπορούμε να σας δώσουμε. Λαμβάνουμε υπόψη μας την παρουσία των βουλευτών, την αίθουσα, τον εξοπλισμό, με μια συγκεκριμένη μέθοδο εργασίας μπορούμε να φτάσουμε σε ένα τελικό νούμερο αφού συμφωνήσουν όλοι ως προς τη διαδικασία. Ναι, προς το παρόν ε, πρέπει να παραμείνουμε σε αυτή την εξήγηση, από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις για την ε, DigiLink. Όχι. Μας μένουν λίγα λεπτά ακόμα και θα ήθελα σε αυτά να επανέλθω σε ένα άλλο πρωταρχικό ερώτημα του κυρίου Μάνκα όσον αφορά αυτήν την ερώτηση που απευθυνόταν σε όλους, σε όλες τις γενικές διευθύνσεις. Αφορά τη συνεργασία μεταξύ των διευθύνσεων. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια από εσάς, αν έχετε κάποια στοιχεία απάντησης. with the other uh, Συνεργασία μεταξύ των διευθύνσεων, συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Νομίζω αυτό ρώτησε ο κύριος Μάνκα. Anyone? Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Κυρία Λίνους; Όχι. Κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά αυτήν την ε, συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων, η Επιτροπή σας εδώ και χρόνια θέλει να στηρίξει αυτήν την θεσμική συνεργασία με σκοπό να κινητοποιηθεί με χαμηλό κόστος το πιο έμπειρο προσωπικό και όλοι από εμάς στο κεφάλαιο 5 διαπιστώνουμε ότι στους διάφορους τομείς δραστηριότητας υπάρχει εντονότατη διαθεσμική συνεργασία η οποία ήδη λειτουργεί Κάποιες φορές γίνεται με πολύ διαρθρωμένο τρόπο, όταν παραδείγματο χάρη έχουμε πρόσβαση σε κάποιους ε, οργανισμούς και θεσμούς οι οποίοι έχουν συσταθεί και ιδρυθεί ε, γι' αυτό το λόγο, όπως τον οργανισμό έψω, όπως ε, τον αρμόδιο φορέα για τις συντάξεις προσωπικού και μελών του Κοινοβουλίου. η Γενική Διεύθυνση law, η tech SAFE έχουν επιτροπές συνεργασίας, κοινέ επιτροπές οι οποίες κυρίως συμμετέχουν σε διαγωνισμούς από κοινού, υποβάλλουν κοινέ προτάσεις. Θα πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί για να μην δημιουργηθούν υπορβολικά μεγάλοι οργανισμοί και φορείς δεν πρέπει να ξεπεράσουμε κάποιο μέγεθος, αλλιώς στο τέλος ο μόνος που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μας θα είναι μια μεγάλη εταιρεία, θα δημιουργήσουμε δηλαδή στρέβλωση του ανταγωνισμού και μονοπωλιακή παροχή υπηρεσίας. Αυτό είναι κάτι που κάθε φορά θα πρέπει να το εξετάζουμε για κάθε δραστηριότητά μας. Ποιο είναι το κριτικό μέγεθος. Ποιο είναι το μέγεθος πέραν το οποίο δεν πρέπει να πάμε. Εγώ στηρίζω την επιθυμία σας για αυτήν την εντονότερη διαθεσμική συνεργασία, αποφεύγοντας περισσότερη γραφειοκρατία όμως. Πολλές φορές ή πολλαπλές τιμολογήσεις ή το γεγονός ότι οι πιστώσεις βρίσκονται στο ένα θεσμικό όργανο και όχι στο άλλο. Χρειάζεται λοιπόν πολλή συνεργασία αλλά εξάλληψη της γραφειοκρατίας. Very much for that. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μάνκα, τρία λεπτά έχουμε ακόμα, τρεις ή λεπτά. Με διερμηνία. Μπορείτε να κάνετε τα τελικά σας σχόλια. Και μία ερώτηση για την οποία φαντάζομαι δεν θα πάρουμε απάντηση. Έχετε τρία λεπτά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γενικούς διευθυντές και γενικές διευθύντριες και για τη δουλειά τους αλλά και για τις παρουσιάσεις τους εδώ σήμερα, πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Στη δική μου έκθεση θα αναφέρω και εγώ το αίτημα περί διαθεσμικής διοργανικής συνεργασίας. Είχα ρωτήσει και στο Προεδρείο γι' αυτό τον Γενικό Γραμματέα Βέλε που παραδέχθηκε ότι περιθώρια βελτίωση υπάρχουν. Και τώρα αναφερθήκατε και εσείς στη μείωση της γραφειοκρατίας για τα τιμολόγια. Άρα, ναι, εδώ μπορούμε κάτι να κάνουμε. Επομένως, θα αναφέρω στην έκθεσή μου τα θέματα αυτά. Πριν 10 χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, εκατομμύρια ευρώ εξοικονομήθηκαν στο πλαίσιο της διοργανικής συνεργασίας, αλλά η βελτίωση είναι μια διαδικασία έναη. Όλοι μπορούμε να βελτιωνόμαστε εσαΐ. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει όλες οι γενικές διευθύνσεις να συνεργάζονται και να αλληλοϊποστηρίζονται. Και αν αυτό οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων, τόσο το καλύτερο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους και προσβλέπω και στην μελλοντική μας συνεργασία. Είμαι πεπισμένος ότι θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Την βλέπω την ε, πρόοδο, είναι αισθητή σε σχέση με τα τελευταία έτη. Και αυτό γιατί υπάρχει φιλοδοξία και προσπάθεια για βελτίωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε κύριε Μάνκα και εξ ονόματός μου ευχαριστίες στις ε, πέντε γενικές διευθύνσεις για τις προσπάθειές τους που ήρθαν εδώ απέναντι στην Επιτροπή μας, αλλά γενικότερα τις προσπάθειες που κάνουν για να μας εξυπηρετούν στην καθημερινή μας ζωή. Ευχαριστώ. Και επόμενη συνδέση Επιτροπής Προπολογισμών την 5η 7 Μαρτίου. Εδώ κυρίσω τη λήξη αυτής της συνεδρίασης και θα συνεχίσουμε και κλεισμένον των θυρών με τη συνεδρίαση των συντονιστών.